So, nach einem langen Pfingstwochenende starten wir jetzt mit unserer Umweltausschusssitzung. Αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Έχω τις εξής ανακοινώσεις. Το σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, καθώς και το 6, θα πρέπει να τα αναβάλουμε. Το 15, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την διερμηνία. Εντάξει. Ολλανδικά. Προς τα Ολλανδικά. Οκ. Λειτουργεί. Ωραία. Λοιπόν, ξαναρχίζω. Καταρχάς, χαιρετίζω συνεδρίαση της Επιτροπής μας, τους παρευρισκόμενους, τα σημεία 6 και 7 ορίζον 2020 και ειδικό πρόγραμμα εφαρμογής του ε, ορίζοντα 2020 αναβάλλονται. Και το 15 είναι η έκθεση Weisgerber θα, το συζήτημα αυτό θα συζητηθεί δημοσίως, όχι και κλεισμένο των θυρών. Το 15 λοιπόν δημοσίως και όχι και κλεισμένο των θυρών. Περνάμε στο σημείο 2. Έχουμε όλες τις γλώσσες στη διάθεσή μας και σήμερα για πρώτη φορά είναι η πρεμιέρα των Κροατικών στην Επιτροπή μας για τους ε, νέους μας συναδέλφους. Δεύτερον, δύο συνάδελφοι παρετήθηκαν από το Κοινοβούλιο, συνάδελφος Ντεμπριν και Ρουμάνα Ρωμάνα Πλάμ, που είναι η νέα Υπουργός Περιβάλλοντος στην ε, Ρουμανία. Οπότε θα την έχουμε απέναντί μας ε, στην άλλη πλευρά της τραπέζης. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για το περιβάλλον στην Ευρώπη και θα ήθελα νομίζω να τη συγχαρώ και προσωπικά και εξ όλων ημών και τη ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην καινούργια της θέση. Οπότε έχουμε δύο νέους αδέλφους εδώ, αναπληρωματικά μέλη. Συνάδελφοι Μιντόρα Σλεβέτη και Ήβαν που αντικαθεστούν τους δύο προηγούμενους. Α, ήρθε... Είναι πίσω από τη συνάδελφο Ιολάν. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Κλειβέτη, μάλιστα το όνομά σας. Καλώς ήρθατε κυρία Κλειβέτη στο Κοινοβούλιο και ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε ορθά. Τρίτη, η ομάδα εργασίας για την υγεία θα συνεδριάσει την Τετάρτη από τις 4 έως τις 6 στην αίθουσα Α5Ε2. Πρόκειται για την ενδιάμεση αναθεώρηση για την στρατηγική της Ένωσης για την Υγεία. Μπορείτε να συμμετάσχετε όλοι. Και τώρα περνάμε στο σημείο ημέρησης διάταξης 3. Ε, έχουμε τον προσκεκλημένο μας κύριο Γιάννους Ποτότσνικ, τον Επίτροπο για θέματα περιβάλλοντος. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Όπως τακτικά κάνουμε και ιδίως εδώ στην Επιτροπή μας, θα έχουμε τρία τμήματα στη συζήτησή μας και έχω ήδη πολλούς συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο αλλά καταρχάς δίνω το λόγο στον Επίτροπο για μια σύντομη εισαγωγή και μετά θα έχετε δυνατότητα να κάνετε ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να λάβουν το λόγο όσο δυνατόν περισσότεροι. Αγαπητέ Γιάννου, έχεις το λόγο. Πέντε λεπτά μια εισαγωγή για το πρώτο θέμα που είναι στην ημερήσια διάταξη σήμερα, που είναι οι νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2013, επικεντρωνόμενοι βεβαίως στην επάρκεια των δημοσιονομικών πόρων. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε να έρθω και να συζητήσω μαζί σας ε, τις εργασίες μας και τα μελλοντικά μας σχέδια. Θα θυμόσαστε πολλοί από εσά ότι στην αρχή της θητείας μου είχα εντοπίσει τρεις τομείς προτεραιότητας που μεταξύ των οποίων ήταν και η δημοσιονομική πόρη, η επάρκειά τους, ήταν και η εφαρμογή και με προσκαλέσατε να έρθω και να σας παρουσιάσω κάθε φορά την πρόοδο που έχουμε επιτύχει. Όσον αφορά αυτό το θέμα λοιπόν το Σεπτέμβριο θέσαμε το πλαίσιο για τις δράσεις που θα έπρεπε να αναλάβουμε έτσι ώστε να υπάρξει βιωσιμότητα μακροπρόθεσμα αλλά και να υπάρχει μια πράσινη όθηση κατά κάποιο τρόπο, ώστε να βγούμε από την τρέχουσα κρίση. Είχαμε την έκθεση και μπράντι την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκε, που έδειξε την πολιτική στήριξη που υπάρχει στην δικιά μας πρόταση. Στήριξη που χρειαζόμαστε και για να προχωρήσουμε παρετέρω. Η έκθεση αυτή που εγκρίθηκε ε, περιλαμβάνει εξαίρετες προτάσεις για, τον, ε, για την πορεία αυτή που πρέπει να ακολουθήσουμε προκειμένου να εφαρμοστούν τα διάφορα μέτρα. Άκουσα μερικέ φορέ τη συζήτηση στην Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα να ε, να λέτε μάλλον ότι ε, δεν προχωράμε αρκετά γρήγορα και δεν προχωράμε στις δράσεις μας όπως θα έπρεπε. Να ξέρετε όμως ε, πως ε, δεν είναι αλήθεια αυτό. Όχι, εμείς προχωράμε σύμφωνα με το φύλλο πορείας πάντα. Το θέμα αυτό της επάρκειας των πόρων αποτέλεσε πάντα εμβληματική η δράση μας από την αρχή της Επιτροπής Μπαρόσο 2. Θέλουμε μια ξεκάθαρη προσέγγιση. Πρώτα απ' όλα να διασφαλίσουμε τους πόρους μας και δεύτερον να ενισχύσουμε τις απαραίτητες αλλαγές που χρειάζονται και τρίτον ε, βελτιωμένη διακυβέρνηση και έλεγχος. Να δώσουμε κίνηση στην ε, ε, κατανάλωση μέσα σε μια εσωτερική αγορά η οποία να έχει πολλά πράσινα προϊόντα. Και το 2013 να ξέρετε ότι θα έχουμε και πρωτοβουλίες για τα βιώσιμα τρόφιμα και τα κτίρια. Η επάρκεια των δημοσιονομικών πόρων είναι μια σαφής έννοια, η οποία καλύπτει και άλλους πόρους, όπως είναι το νερό. Ε, Φέτο ακόμα θα υποβάλουμε ανακοίνωση για την προστασία των υδάτινων πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης στα τέλη του 2013 θα υπάρξει και μια πλήρης αναθεώρηση της πολιτικής μας όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, βασιζόμενη στις, στην τελευταία συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Γενέβη προκειμένου να τροποποιηθεί το πρωτόκολλο Βέντεμπορκ. Όμως, βέβαια, η επάρκεια των πόρων είναι κάτι πολύ σημαντικό ε, στα πλαίσια της ατζέντα μας και σημαίνει ότι θέλουμε να ληφθεί υπόψη και στα πλαίσια άλλων πολιτικών και στην εφαρμογή της στρατηγικής μας έτσι όπως αυτή οθετήθηκε πέρυσι για το 2020. Να ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό να φέρουμε σε πέρα τις ε, υποχρεώσεις που αναλάβαμε, να συμπληρώσουμε το πλαίσιο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δουλεύουμε επίσης και βάσει ενός ε, μέσου για διάφορα σπάνια είδη. Επίσης συνεχίζουμε το έργο μας για την εφαρμογή της νομοθεσίας όσον αφορά τις χημικές ουσίες αλλά εγκρίνοντας ε, πολιτική και νομοθεσία για τις πολιτικές μας είναι το πρώτο βήμα. Για να αποφεληθούμε από τα μέτρα αυτά, τα τωρινά και τα μελλοντικά σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται και σωστά εφαρμογή τους. Περιμένω την δικιά σας ε, λοιπόν άποψη όσον αφορά το άγγραφο που ενέκρινε η Επιτροπή το Μάρτιο για την εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων, κάτι που θα συμπληρωθεί και με τα επόμενα μέτρα από την οδηγία αντικτύπου, όπου θέλουμε να διασφαλίσουμε μια πιο συνεπή εφαρμογή των αρχών που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση του περιβάλλοντος. Η προσέγγιση αυτή τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ό,τι αφορά τους άλλους γίνεται και δικιά μας δουλειά. Δηλαδή στην εφαρμογή της πολιτικής μας ασχολούμαστε με την ενέργεια, τις μεταφορές, την ε, συνοχή στη γεωργική μας πολιτική, την αναλία, αλλά και τις εξωτερικές μας πολιτικές. Οι συζητήσεις που γίνονται βάσει της πρότασης της Επιτροπής, βάσει του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, είναι κάτι που αποτελεί σημαντική δοκιμή, προκειμένου να δούμε αν αυτέ τι αρχέ μπορούμε να τι εφαρμόσουμε και σε άλλε πολιτικέ. Ελπίζω ότι μπορώ να βασιστώ στα μέλη τη Επιτροπή αυτή, προκειμένου η επάρκεια αυτή πόρων να αποτελέσει βασικό στοιχείο ε, στον πυρήνα της δουλειάς που κάνουν και άλλες επιτροπές γεωργίας, ε, μεταφορών, αλίας κλπ. κλπ. Θα συνεχίσουμε εξάλλου και το διάλογο με τα κράτη-μέλη για θέματα όπως είναι το θέμα του πρασινίσματος των ε, φορολογικών συστημάτων, των επιδοτήσεων και της ανάπτυξης που πρέπει να βασίζεται σε πράσινα μέτρα. Είναι ο καλύτερος τρόπος, πιστεύουμε, για να γίνεται η συζήτηση αυτή και ε, να ληφθεί υπόψη και στα πλαίσια της πολιτικής για την οικονομική διακυβέρνηση και τη στρατηγική 2020. Όπω ξέρετε, οι συζητήσεις αυτές ε, γίνονται τώρα. Αύριο θα τι συζητήσουμε στι συνεδρίε τη Επιτροπή. Δείκτε επίση, και στόχοι είναι και αυτά πράγματα που αποτελούν προτεραιότητα για μα. Έχουμε ξεκινήσει φέτο την ε, διαδικασία πέρα από την πλατφόρμα αυτή για την επάρκεια πόρων που θα αποτελέσουν τη βάση για την πολιτική μα για το 2013. Τέλος, Φέτος ακόμα στα τέλη της χρονιάς θα έχουμε πρόταση για ένα νέο πλαίσιο για την πολιτική περιβάλλοντος που να βασίζεται στο πρόγραμμα πλαίσιο για το περιβάλλον. Εμείς χαιρόμαστε για τη δουλειά που έχει κάνει η δικιά σας επιτροπή, την έκθεση Γιολάινεν και θέλω την στήριξή σας προκειμένου να ετοιμάσουμε ένα νέο σχέδιο που να αντιμετωπίζει τις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις και να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης για το 2020 που να βασίζονται στην ανάπτυξη και την ευημερία. Όσο προχωράμε χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ μας προκειμένου όλοι αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι να γίνουν πραγματικότητα με απτά αποτελέσματα και πλεονεκτήματα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ξέρω ότι η εφαρμογή είναι στο τρίτο σημείο και το ρίο και το... τα ύδατα είναι στο δεύτερο σημείο, αλλά όταν μιλάμε για την επάρκεια πόρων δεν είναι δυνατόν να μην μιλήσουμε και για όλα αυτά συγχρόνω. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Επίτροπε Ποτότσνικ για αυτή την ε, σύντομη επισκόπηση για όλα όσα σχεδιάζεται Εφόσον πρόκειται για νομοθετικές εκθέσεις, για νομοθεσία, η προθεσμία για το Κοινοβούλιο είναι ο Μάρτιος του 2013. Δηλαδή, όποιες προτάσεις. Δεν, δεν υπάρχει διερμηνία. Α. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση εφόσον πρόκειται για νομοθεσία, για νομοθετικές εκθέσεις εδώ στο Κοινοβούλιο, η προθεσμία είναι Μάρτιος του 2013. Γιατί οποιασδήποτε προτάσεις υποβληθούν ε, από την Κομισιόν αργότερα, δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα να τα αντιμετωπίσει το Κοινοβούλιο στην νομοθετική περίοδο, γιατί ήδη το Μάρτιο του 2013 Σιγά σιγά θα μπούμε στην προεκλογική περίοδο. Και από τον Απρίλιο δεν θα γίνει πια καμία συνεδρίαση. Σας παρακαλώ λοιπόν όλες τις νομοθετικές προτάσεις να τις κάνετε πριν από το Μάρτιο του 2013 για να έχουμε τη δυνατότητα κατά αυτή την νομοθετική περίοδο να ε, εφαρμόσουμε αυτές τις προτάσεις. Μιλήσατε για την αποτελεσματική χρήση πόρων. Το έχουμε ήδη συζητήσει και προηγουμένω. Νομίζω ότι κάναμε μια ιδιαίτερα χρήσιμη συζήτηση στα πλαίσια τη έκθεση Κερμπράντι. Συνέβαλαν, ε, μίλησαν δηλαδή πάνω από 50 άτομα. Αυτό αποδεικνύει ότι το θέμα σε πολύ μεγάλο βαθμό μα ενδιαφέρει. Λοιπόν, να μην πω πολλά. Πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο. Πρώτο, ο Ρίχαρτ Τζέιμπα από πλευρά του ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. οι συζητήσεις που κάνουμε για το περιβάλλον πάντα είναι έντονες και αυτό είναι λογικό. Καταρχάς ευχαριστώ τον Επίτροπο και το συγχαίρω για την τελευταία πράσινη εβδομάδα η οποία πήγε πολύ καλά. Νομίζω ήταν μια θαυμάσια πρωτοβουλία να δείξει στους πολίτες μας τι κάνει η Ευρώπη για το περιβάλλον. Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση. Όχι μόνο να έχουμε σωστούς κανόνες, αλλά να ευαισθητοποιούμε και την κοινή γνώμη. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα για την ε, περιβαλλοντική νομοθεσία. Υπάρχουν πολύ μεγάλες ανισότητες στην εφαρμογή. του. ανέφερε και ο Επίτροπος για το πρόγραμμα εργασίας ε, της Κομισιόν για αυτή τη θητεία. Αλλά δεν έχουν σημειωθεί θεαματικές πρόοδοι, πιστεύω, στον τομέα αυτό. Για τα ύδατα και την ατμόσφαιρα όπως ξέρετε για την ατμόσφαιρα είπατε ότι του χρόνου θα υπάρξει μια αναθεώρηση της ποιότητας, ε, της, ε, των ε, ενεργειών που κάνουμε για την ποιότητα του αέρα. Αλλά παρόλα όσα έχουμε κάνει εξακολουθεί να είναι κακή η ποιότητα του, του ατμοσφαιρικού αέρα παρόλες τις προσπάθειές μας, παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας, παρά τους περιορισμούς για την θέρμανση. Παρόλα αυτά δεν επιτυχάνουμε τους στόχους μας. Απέχουμε πολύ. Όπως είπα, έχουν γίνει πολλές αιτήσει για να βελτιωθεί η κατάστασή μας ε, στον τομέα αυτό, ακόμη και έξω από την Ευρώπη. Πρέπει να επιλέξουμε λοιπόν μια προσέγγιση που να αντιμετωπίσει αυτή την ειδική κατάσταση. Δηλαδή να τηρούμε τις οριακές τιμές. Διότι αυτή τη στιγμή δεν το καταφέρνουμε. Το ίδιο και στα ύδατα. Έχουμε την προτεραιότητα για αυτές τις ε, ενώσεις προτεραιότητας, αλλά και εδώ θέτουμε κάποιες τιμές κατοφλίου, αλλά ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο τα κράτη-μέλη να κάνουν πολύ δαπανηρές επενδύσεις για καταστάσεις ε, κατεργασίας των αποβλήτων και για χρόνια δεν επιτυχάνουμε αυτές τις τιμές, οπότε είναι πρόβλημα. Δηλαδή το μήνυμα που στέλνουμε είναι ότι παρά την πλήρη πολιτική μας βούληση και παρά τις τεράστιες επενδύσεις δεν επιτυχάνουν τα κράτη-μέλη τους στόχους και αυτό είναι απογοητευτικό. Πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε κάποια άλλη αντιμετώπιση, να έχουμε άλλη διαδικασία εγκρίσεων, να έχουμε συνδυασμό εγκρίσεων, να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά τη βιομηχανία και επίσης θα παρακαλούσα τον Επίτροπο, επειδή έχουμε ακόμα ένα χρόνο, προσπαθούμε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε συγκεκριμένα τα κράτη-μέλη. Δεν θέλουμε να επιχειρήσουμε εντελώ νέες προσεγγίσεις, απλώς να βελτιώσουμε την εφαρμογή. Έτσι θα κάναμε κάτι συγκεκριμένο για τους Ευρωπαίους ε, πολίτες. Γιολάινεν. Κύριε Επίτροπε, εάν ε, γίνει τόσο γρήγορα και η εφαρμογή της νομοθεσίας όσο γρήγορη ήταν η παρουσίασή σας, τότε θα επιτύχουμε πολλά πράγματα. Πραγματικά, σε πέντε λεπτά τα, τα είπατε όλα. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι νόμους μπορούμε, τι νομοθετήματα μπορούμε να περιμένουμε ότι θα μας έχετε υποβάλει μέχρι το Μάρτιο του 2013 για την αποτελεσματική χρήση πόρων για παράδειγμα ή θα πρέπει να αναβληθεί για την επόμενη θητεία το θέμα αυτό. Και επίσης, πώς είναι η σύνδεση μεταξύ του 7ου περιβαλλοντικού προγράμματο, του προγράμματο ε, ε, αποτελεσματική χρήση των πόρων και του προγράμματο βιωσιμότητα. Πώ προχωράνε από, μαζί, από κοινού τα θέματα αυτά για το τρίτο, στρατηγική βιωσιμότητα. Δεν βλέπω να προχωράει πολύ. Έχει βραδιπορήσει, θα υπάρξει νέα όθηση, νέα δυναμική για το θέμα αυτό. Πώς συνδυάζονται αυτές οι τρεις δράσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια τέθηκε και ένα ερώτημα προς τα, προς κράτη-μέλη. Αν έχουν προγράμματα δράσης για τους πόρους, για την ε, προστασία του κλίματος, έχουμε τις ενέργειες μετριασμού. Υπάρχουν παρόμοια σχέδια στα κράτη-μέλη για την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Από ό,τι ξέρω, μεθαύριο η γερμανική κυβέρνηση θα παρουσιάσει το πρόγραμμα δράσης της για την αποτελεσματική χρήση πόρων. Θα θέλαμε να το έχουν όλα τα κράτη-μέλη αυτό, για να έχουμε μια συνολική εικόνα και να μπορούμε να μετράμε από χρόνο σε χρόνο τι πρόοδος έχει σημειωθεί. Δύο ακόμη για τα νομοθετήματα. Ο θόρυβος, σημαντικό θέμα. Για το θέμα αυτό θα υπάρξει βελτίωση της νομοθετικής εργασίας. Ο κύριος Ζέμπερ αναφέρθηκε στον ατμοσφαιρικό αέρα. Αλλά αυτός είναι ο εξωτερικός αέρας. Οι περισσότεροι τον περισσότερο χρόνο τον περνάνε σε κλειστούς χώρους. Και εδώ έχουμε προβλήματα. Υπάρχει πρόγραμμα για τη βελτίωση του αέρα εντός των κτηρίων όπου ζουν και εργάζονται ε, οι πολίτες μας. Ευχαριστώ. Chris Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναφερθήκατε στην νομοθεσία. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε όμως προσεκτικοί έτσι ώστε να μην ασχοληθούμε μόνο με τα θέματα πρώτης ανάγνωσης και αυτό για πολλούς λόγους. Δηλαδή να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα των συμβιβασμών της πρώτης ανάγνωσης που ενδεχομένως δεν θα φτάσουν τελικά σε ένα ικανοποιητικό ε, αποτέλεσμα και στο τέλος μάλιστα και το Συμβούλιο θα μας θεωρήσει δεδομένους. και επομένως ε, δεν θα θεωρήσει ότι πρέπει να συζητιέται και πολύ. Ε, λοιπόν, ε, είδαμε κάποια έγγραφα, δεν είδαμε όμως πολύ ουσία που να αποδεικνύει ότι η Κομισιόν τελικά επιτυγχάνει περισσότερα πράγματα ε, ε όσον αφορά την εφαρμογή. Ελπίζω να έχετε τη δυνατότητα να μας αποδείξετε το αντίθετο. Θα σας δώσω κάποιο παράδειγμα. Κατά την άποψή μου, υπάρχει ένα έγγραφο. 2000. 2006... Um, από το 2006 απαιτείται όλα τα κράτη-μέλη να καλύπτουν το 85% ε, του κομματιού του κάθε χήματος που ανακυκλώνουμε και από το 2015 αυτό πρέπει να αυξηθεί στο 95%. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, οι περισσότερες ε, χώρες ε, μέλη καλύπτουν το 85% τώρα. Και άλλες κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά δεν υπάρχει πίεση πάνω σε αυτές, ώστε να ανταποκριθούν στις νόμιμες απαιτήσει και απλώς προσπαθούν να πιέσουν τους εαυτούς τους έτσι ώστε να ε, προσαρμοστούν όσο γίνεται καλύτερα. Τώρα ε, υπάρχουν χώρες οι οποίες ε, προσπαθούν ε, να, προσπαθούμε μάλλον τώρα να έχουμε ένα επίπεδο για όλη την Ευρώπη έτσι ώστε να μην υπάρχει εσωτερικό συνταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά θα πρέπει η Κομισιόν, οφείλει δηλαδή, να πιέσει τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να έχουμε πραγματική μείωση και έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα από ό,τι φαίνεται και από, ό,τι, από βλέπω το ύφο σας, δεν φαίνεται να το θεωρήσατε πάρα πολύ σημαντικό ε, το ζήτημα αυτό. Ε, και ε, γι' αυτό λοιπόν σας ρωτώ ποια είναι τα μέτρα παραβάση, συγκεκριμένες πράξεις οι οποίες προτίθεστε να αναλάβετε έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι προτάσεις της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ε, και επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έμαθες ότι η φυσιολογική διαδικασία ε, έχει δύο αναγνώσεις. Σύμπας. Επόμενος ομιλητής. Ε, Μπέστα Ευχαριστώ πολύ. Αρχηγέ. Και ευχαριστώ και εσάς, Επίτροπε Ποτότσνικ, που ήρθατε εδώ. Όντω ε, πιστεύω ότι και με την έκθεση που εγκρίναμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια ε, δείχνουμε σαφώ ε, ποιο είναι ο προσανατολισμό που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Αλλά τώρα βεβαίω πρέπει να ακολουθήσουν και οι πράξει, η εφαρμογή. Γιατί βεβαίω έχουμε ένα όραμα με το οποίο συμφωνούμε όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Θέλουμε να υπάρξουν διασυνδέσει και γέφυρε ανάμεσα σε όλου του εμπλεκόμενου, πολιτικέ ομάδε του Κοινοβουλίου κτλ. Αλλά τώρα θα πρέπει πρέπει να φτάσουμε στις πράξεις και αυτό άλλωστε αποζητούν όλοι, αυτό είναι και το ζητούμενο. Θα ήθελα να επιστρέψω την προσοχή σας επί τριών σημείων, επί των οποίων θα θέλαμε κάποιες αποσαφηνήσει. Πρώτον, Βεβαίως η οδηγία ε, αναφέρθηκε και στην έκθεσή μας και εκεί ρητά ε, είπαμε ότι θα πρέπει να διευρυνθεί η οδηγία ε, και θα πρέπει να αναφέρεται και σε μη ενεργειακά προϊόντα και θα πρέπει βεβαίως να γίνει προσπάθεια να ενισχυθεί η ενεργειακή απόδοση. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε πότε μπορούμε να περιμένουμε κάποια διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και επίσης και ιδίως ε, αυτό, αυτή η δέσμη θα φτάσει πριν από τον Μάρτιο του επόμενου έτους. Δεύτερον, βιομάζα. Δέστε λίγο πώς μας απασχολεί, πώς αντιμετωπίζουμε τη βιομάζα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ε, με την συγχρηματοδότηση η οποία ήδη από μόνη της είναι ανεπιτυχής και ανεπαρκής σε ανεπαρκής ε, υποδομές. Εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξουν και κάποια κριτήρια υφορίας. Υπάρχει μια συζήτηση βέβαια που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή αλλά πότε θα έχουμε απτά συγκεκριμένα και ε, ε, και φιλόδοξα κριτήρια αηφορίας όσον αφορά την βιομάζα ε, έτσι ώστε να αποφύγουμε συγχρηματοδότηση ανεπιτυχών υποδομών. Τρίτον, είμαι λίγο από είμαι λίγο έτσι απογοητευμένος γιατί στην ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ βλέπουμε κάποια, σχετικά υπάρχει πρόοδο όσον αφορά το πρασίνισμα και τα λοιπά, αλλά πιστεύω ότι χάνουμε και κάποιες ευκαιρίες. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ε, ε, η γενική σας διεύθυνση ε, συζητάει, δουλεύει πάνω σε ένα έγγραφο ε, σχετικά με τα φωσφορικά. Ε, ξέρουμε ότι γίνεται κάποια δουλειά, αλλά θέλουμε να δούμε εάν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας για τα φωσφορικά και με άλλες γενικές διευθύνσεις, Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας ας πούμε, έτσι ώστε ε, να μην κάνουμε εισαγωγές από το Μαρόκο και τελικά να, να τα ρίχνουμε στον ωκεανό, να τα ποντίζουμε τα απόβλητα των φωσφορικών αλάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ähm, Ευχαριστώ. Θα μιλήσω δανέζικα καλύτερα. Για τα νοικοκυριά, τα ιδιωτικά δηλαδή νοικοκυριά. Με όλη αυτή την νομοθεσία, πώς νομίζετε ότι τα ιδιωτικά νοικοκυριά θα μπορέσουν να εφαρμόσουν όλα αυτά Πώς δηλαδή όλα αυτά τα μέτρα θα φτάσουν ατομικά στον κάθε πολίτη. Έχουμε διάφορα έγγραφα εδώ και πολλές φορές είναι καλό να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο και να μην φτάνουν στον κόσμο γιατί ο κόσμος είναι αυτός τελικά που πρέπει να αλλάξει τον κόσμο. Άρα πρέπει να μπορεί. Ο κόσμος δηλαδή ο καθημερινός, ε, τα νοικοκυριά. Ενέργεια, φωτισμός, ε, μόνωση, ε, για να αποφεύγουμε τη ζέστη, το κρύο, ε, τα διάφορα πλαίσια. Και... Πάλι υπάρχει πρόβλημα με την διερμηνία, λέει ο πρόεδρος, από τα, ε, μάλλον προς τα γαλλικά. Προτιμάτε να μιλήσω γερμανικά, λέει η ομιλήτρια. Man for eksempel øh, PR, television eller... Έλεγα λοιπόν, συνεχίζει η ομιλήτρια, έχουμε την τηλεόραση και άλλους τρόπους να φτάσει το μήνυμα στους ανθρώπους, στον κόσμο, ώστε να καταλάβει ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στις καθημερινές μας συνήθειες και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους ενεργειακούς πόρους στην καθημερινή ζωή. Αναφερθήκαμε πριν στο είδωρ, την ατμοσφαιρική ρήπανση. Τι γίνεται όμως με τα απόβλητα από τα φάρμακα που φτάχνουν στο νερό. Και το νερό αυτό φτάνει όχι μόνο στη Γεωργία, αλλά και στην Αλία. Οπότε ρωτάω, τι κάνουμε γι' αυτά. Γνωρίζουμε αρκετά καλά τι γίνεται με τα απόβλητα από την γεωργία, αλλά από τις υδατοκαλλιέργειες έχουμε εκεί κάποιο στοιχείο. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ. Ρώσο, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Χαίρομαι κύριε Επίτροπε γιατί είστε εδώ, γιατί θέλω να σας ρωτήσω πώς ε, συμφιλιώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό αυτό, αυτή την ακριβή μάχη για το διοξίδιο του άνθρακος από τη μία πλευρά με την απόλυτη με την απόλυτη αδιαφορία ε, για την ε, ύπαρξη χωματερών όπου αποβάλλονται ε, ένα σωρό καρκινογόνες ουσίες κρυβόμενος πίσω από το σλόγγαν «Μα για αυτά που είναι υπεύθυνα τα κράτη-μέλη». Μα για αυτα ειναι ότι αυτές οι χωματερές είναι γεμάτες με καρκινογόνες και και τερατογόνες ουσίες, είναι γεμάτες δηλητήριο. Και τι λέτε εσείς, εντάξει, λέτε ότι πρέπει να πληρώνονται ε, τα ποσοστά, τα οποία είναι όλο και πιο ακριβά και ο συνάδελφος σας ο κ. Σαλμούνια λέει και παραθέτω, εάν οι παραγωγές περνάνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτες χώρες οι οποίες έχουν λιγότερο αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία, αυτό θα μπορούσε να δυναμητήσει τον ε, στόχο μας για συνολική μείωση των ε, αερίων του θερμοκηπίου. Επομένως, θα πρέπει να δίνονται επιδοτήσεις έως και 80% των δαπανών των ε, επιχειρήσεων μεταξύ του 13 και 15 ε, ποσοστό το οποίο θα κατεβεί στο 75% μέχρι το 2020. Ποιος θα πληρώσει θα πληρώσουν με ένα σχήμα κρατικών επιδοτήσεων τα κράτη-μέλη ε, ε, συνεπικουρούμενοι από την ε, βιομηχανία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για αγορά ποσοστών διοξιδίου του άνθρακα μετά μέχρι 85% του κόστους της ενέργειας για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις και βιομηχανίες θα πληρώσουν όλοι οι Μετά όμως λέτε, α καλά εμείς όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τα αποβλητά λεφτά σα, θα πληρώσετε για να αγοράσετε, αλλά το τι θα κάνετε μετά είναι δικό σας θέμα. Τι θα γίνει κύριε Επίτροπε, Υπάρχουν ε, ε, χώρες και η δικιά μου η χώρα είναι γεμάτη στο υπέδαφος της με καρκινογόνες ε, ουσίες. Ούτε το κράτος, ούτε η περιφέρεια, ούτε ο Δήμος, ούτε η κοινότητα δεν προσπαθεί να εξηγιάνει το υπέδαφος. Δηλαδή εσείς τι μας λέτε, μας λέτε ότι καθίστε εκεί στην ησυχία σας και, και πεθάνετε σιγά σιγά ή μας λέτε ότι εδώ θα έχουμε μπουκαλάκια νερού ε, που θα τα γεμίζουμε με διοξίδιο του άνθρακο και θα, τα, ε, θα τη ζωή μας τελικά. Έκλεισε ο πρώτος γύρος ε, ομιλητών. Μιλήσαμε για αποδοτικότητα των πόρων, προγράμματα δράσης. Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε τους στόχους μας, αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε ένα εθελοντικό σύστημα με τη βιομηχανία, που όμως δεν απέδωσε. Και και αν η Επιτροπή θέλει να, θέλει να, αναλυφθεί το εξωτερικό κόστος από εσωτερικούς φορείς, όπως τον τομέα της, ε, των μεταφορών, αν θέλει να το εφαρμόσει, να εφαρμόσει αυτή την αρχή και στον τομέα της, ε, του περιβάλλοντος, και αυτό ζήτησε μία έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής μας, θα θέλαμε η Επιτροπή να μας πει τι εννοεί, πώς θα γίνει η χρηματοδότηση, να κάνουμε τη συζήτηση για το εάν θα γίνει μέσω φορολόγησης. Αν πραγματικά θέλουμε κάτι να αλλάξουμε για τα ύδατα και για άλλες ουσίες, θα πρέπει όλες αυτές οι ουσίες να έχουν κάποια τιμή. Όλα αυτά πληρώνονται τώρα από τον προπολογισμό υγείας και από τους φόρους. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε διαφορετική προσέγγιση. Παρακαλώ κύριε Επιτρόπε. αρκετά μακρύς κατάλογος. Αν χρειαστεί να εξηγήσω ορισμένα από τα θέματα για τον διαρθρωμένο διάλογο υπό τα σημεία 2 και 3 μπορεί και να μπερδευτώ, αλλά ο Ρίχαρτ πρώτος έθεσε τα θέματα εφαρμογής για το σημείο 3. Οπωσδήποτε σημαντικό θέμα. Είπατε σε πολλές περιπτώσεις δεν βλέπουμε συγκεκριμένες προόδους. Αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχουν όμως ε, σοβαροί λόγοι για την ε, μη εφαρμογή και οι διαφορές μεταξύ 100 μελών είναι τεράστιες. Έχουμε τώρα μία νέα προσέγγιση ε, εξέτασης, επιτήρησης της εφαρμογής με τη νέα μας ανακοίνωση, όπου μιλάμε για τις ρίζες του προβλήματος. Δύο είναι τα βασικά προβλήματα στην Ευρώπη. Το πρώτο είναι ότι οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τις κυβερνήσεις τους και το δεύτερο είναι ότι οι κυβερνήσεις δεν εμπιστεύονται μία την άλλη. Και αυτό δημιουργεί τα κυριότερα προβλήματα της εφαρμογής, που πρέπει όλοι μαζί να τα αντιμετωπίσουμε. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε μια πιο συστηματική προσέγγιση της γνώσης. Διότι πολλές φορές αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό ad hoc. Και το δεύτερο, να αυξήσουμε τη δυνατότητα των κρατών μελών να αποκτήσουν ε, παρόμοια συστήματα και όλοι οι θεσμοί, οι επιθεωρητές, οι δικαστικοί, οι κυβερνήσεις να δρουν με συγκρίσιμο τρόπο. Και αυτό θα πείσει και τους πολίτες ότι οι κυβερνήσεις τους, τα θεσμικά τους όργανα μπορούν να κάνουν αυτά που υπόσχονται. Αυτά τα θέματα θέλαμε να τονίσουμε μέσω της ανακοίνωσης. Φυσικά ίσως ε, να προτιμούσαμε αυτή η ευαισθητοποίηση να γίνει περισσότερο μέσω του νομοθετικού προγράμματος. Μπορούμε βέβαια να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε κατά περίπτωση τις παραβάσεις, όπως είπε και ο Κρίς. Αλλά, όπως ξέρετε, θα συζητήσουμε για την διαδικασία παραβάσεων ε, στην ε, πολιτική μας για τον ατμοσφαιρικό αέρα. Βεβαίω πρέπει να θέτουμε προτεραιότητε όσον αφορά την εφαρμογή. Βεβαίω. Ναι, μεν πρέπει να ε, τιμωρηθούν όλοι όσοι παραβιάζουν τον νόμο, αλλά όταν έχουμε εκατοντάδε παραβιάσει, πρέπει να θέσουμε κάποιε προτεραιότητε. Ποιε θα αντιμετωπίσουμε πρώτα, αυτέ που έχουν ε, σοβαρότερε επιπτώσει, αυτέ που γίνονται εδώ και περισσότερο καιρό, που επηρεάζουν μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, δεν ξέρω. Γιατί ξέρετε δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα την ίδια στιγμή. Υπερβαίνει τις δυνατότητέ μας. Το αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα με μεγάλη σοβαρότητα. Αλλά κοιτάξτε, έχουμε 470 άτομα που εργάζονται όλοι πάρα πολύ σκληρά. Κάνουν ό,τι μπορούν. Αλλά κάθε μέρα μας ζητάνε να κλείσουμε κάποια ζητήματα και δεν είναι πρόφαση αυτό. Θα θέλαμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα, αλλά αντικειμενικά είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο παράλληλα να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα με την ίδια αποφασιστικότητα. Ρωτήσατε τι θα γίνει του χρόνου. Βεβαίω, μας ενδιαφέρει η αναθεώρηση της πολιτικής για τον ατμοσφαιρικό αέρα. Μόλις σήμερα είπα ότι η συζήτηση θα είναι πολύ δύσκολη, η συζήτηση για το θέμα αυτό, διότι η πολιτική για τον ατμοσφαιρικό αέρα δεν είναι εύκολο θέμα. Για να το αντιμετωπίσουμε πρέπει να βρούμε τη ρίζα του προβλήματος, δηλαδή να δούμε πώς εργαζόμαστε σε άλλους τομείς και να συνδυάσουμε τις προσπαθειές μας για να δώσουμε αποτελεσματικές λύσεις. Όταν συζητήσαμε το πρωτόκολλο του Γκέτεμποργκ υπήρχαν μεγάλες δυσχέρειες και ευτυχώς δεσμεύτηκαν τα κράτη-μέλη για κάποιους φιλόδοξους στόχους που συνδυάζονται με το 2020. Θα υπάρξει μια αναθεώρηση επίσης και της οδηγίας ΝΕΚ. Όπως ξέρετε έχει αναβληθεί επανειλημμένα γιατί και αυτό συνδέεται με τις σοβαρές προσπάθειες πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη. Αλλά έχουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σημαντικά στοιχεία. Είναι ότι αυτό που θίγει ουσιοδός την ανθρώπινη υγεία είναι η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Συνδέεται με μια σειρά από ασθένειες, άσθμα και παρόμοιες, μέχρι τη μείωση του μέσου όρου ζωής της πόλης ε, σε σχέση με την Ήπεθρο. Πρέπει λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε. Το άλλο θέμα που πρέπει οπωσδήποτε να είναι στο κέντρο της προσοχής μας είναι να ξεκινήσει αυτή η μεταβατική πλατφόρμα για την αποδοτικότητα των πόρων. Έχω υψηλές προσδοκίες για το θέμα αυτό. Με αυτόν τον τρόπο θα ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη για το θέμα αυτό και τις κυβερνήσεις, γιατί δεν υπάρχει επαρκής συνειδητοποίηση για το θέμα αυτό, θα υπάρξει πολιτική βούληση για την εφαρμογή, αλλά και για τον καθορισμό στόχων και δικτών, γιατί είναι ουσιώδης, θεμελιώδης. Θα σας διαβάσω κατόπιν ε, ορισμένα στοιχεία από το Παγκόσμιο Συμβούλιο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη εν ώψη του Ρίο. Είναι 200 εταιρείε από όλο τον κόσμο με τζίρο πάνω από 7-3. 7 στόχοι. Να έχουμε συγκεκριμένους στόχους, να ενημερώνουμε, να ρυθμίζουμε, να έχουμε προϋπολογισμό, να συντονίζουμε, να ε, επενδύουμε και να ελέγχουμε. Αν θέλουμε να ακούσουμε τις συμβουλές τους, πρέπει ακριβώς να τις εντάξουμε σε αυτήν τη νέα πλατφόρμα για την αποδοτικότητα. Τη, χρειαζόμα, τη χρειαζόμαστε απεγνωσμένα και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να υπάρξει σαφέστερη εφαρμογή στο μέλλον. Για τον ΝΑΙΣ, είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα. το, η έκθεση Συγγνώμη για τον θόρυβο, για το θόρυβο υποθέτουμε. Ε, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή της οδηγίας πρόσφατα, ε, μάλλον ε, προσεχώς. Θα ξεκινήσουμε την ε, διαδικασία αναθεώρησης ε, του θέματος αυτού και θα προσπαθήσουμε να υπάρξουν κοινέ μέθοδοι για να αποτιμήσουμε και να μετρήσουμε επίπεδα θορύβου σε όλη την Ένωση. Ήδη λοιπόν οδεύουμε αυτή την οδό, πιέζουμε για να εφαρμοστούν περισσότερο τα μέτρα. Για την εφαρμογή ήδη μίλησα, οικολογικό σχεδιασμός, θα υπάρξει θέση για την επέκταση του τομέα εφαρμογής μέχρι το τέλος του 12. Κάναμε μια μελέτη αποτίμησης και τα συμπεράσματα λένε ότι εάν επιχειρήσουμε να επεκτείνουμε το παιδί εφαρμογή θα ήταν λίγο πρόωρο, ενώ βεβαίω μπορεί να έχει σημαντική οικολογική επίπτωση η επέκταση, αλλά οι μέθοδοι δεν είναι ακόμη στη διάθεσή μας και θα υπήρχε υψηλός κίνδυνος να μην υπάρξει συμμόρφωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν άσκοπη η εργασία μας ως τώρα, αλλά πρέπει να αναπτύξουμε νέες μεθόδους ελέγχου του ε, περιβαλλοντικού ίχνους και θέλουμε να προωθήσουμε και συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα για την σήμανση. Όλα αυτά θα είναι σημαντικά. Πιστεύω απόλυτα στον οικολογικό σχεδιασμό. Θα πρέπει να περάσει και πέρα από την ενέργεια, να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του, αλλά πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο που να είμαστε σίγουροι ότι βαδίζουμε σωστά, σίγουροι ότι μπορούμε πραγματικά να τα εφαρμόσουμε όσο αποφασίζουμε. Μιλήσατε για θέματα βιομάζας. Είναι απόλυτα αναγκαίο να μην λαμβάνουμε λανθασμένες αποφάσεις. Γιατί τότε κλείνει ένα θέμα με λάθος τρόπο. Δεν λαμβάνουμε δηλαδή υπόψη τις παρενέργειες που μπορεί να υπάρξουν σε άλλους τομείς λόγω εφαρμογής κάποιου μέτρου. Και ξαφνικά προκύπτουν ε, προβλήματα που δεν τα είχαμε προβλέψει. Άρα να μην δαπανίσουμε ασκόπως ε, τους πόρους μας. Για τη βιομάζα ακούσαμε βεβαίως ε, τις απόψεις εμπειρογνωμόνων. Υπάρχουν ε, αποκλίνουσες, πολύ αποκλίνουσες απόψεις. Πιστεύουμε βεβαίως ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Η σημερινή κατάσταση δεν επαρκεί, αλλά τι περαιτέρω μέτρα. Εγώ πιστεύω ότι οποτεδήποτε κάνουμε τέτοιες ε, αναθεωρήσεις, επισκοπήσεις, να μην ξεχνάμε το εξής. Γιατί θέλουμε τη βιομάζα και γιατί υιοθετήσαμε όλες τις πολιτικές ανανεωσίμων ενεργειών. Γιατί υπάρχει κίνδυνος κλιματικής αλλαγής και άρα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Να αντιμετωπιστούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Άρα να το λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό όταν συζητάμε τα θέματα αυτά. Είναι απόλυτα αναγκαίο να μην ξεχάσουμε το στόχο μας. Επειδή τώρα επενδύσαμε τόσο πολλά, αν ξεχάσουμε Ποιο είναι ο βασικός λόγος που αρχίσαμε να εφαρμόζουμε αυτές τις πολιτικές, τότε θα πέσουμε έξω. Θα χάσουμε το στόχο από το οπτικό μας πεδίο. Για τη βιομάζα λοιπόν και για τον κύκλο των τροφίμων και τις ε, φωσφορικές ουσίες. Μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρξει μια ανακοίνωση. Κουίν, Ταγιάννη και εγώ θα συνεργαστούμε εδώ λοιπόν μπορούμε να συνδυάσουμε την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Τώρα, για την αποδοτικότητα και πάλι. Για τις φωσφορούχες ουσίες είπα. Αλλά για την αποδοτικότητα των πόρων είπα ότι προετοιμάζουμε για του χρόνου δύο έγγραφα για δύο τομείς που θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα. Η κινητικότητα που αναφέρθηκε και στη Λευκή Βίβλο, τα τρόφιμα, βεβαίω συμπεριλαμβάνονται και το τρίτο, τα κτίρια. Και εδώ θα υπάρξει ένα κείμενο που είναι συνέχεια όλων όσων έχουμε ήδη πει για την αποδοτικότητα με πολύ πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Για την διάδοση βεβαίως. Είναι θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Ο εφιάλτης μου είναι ότι πάντα όταν μιλάμε για την αποδοτικότητα όλοι μου οι συνάδελφοι και διάφοροι που ασχολούνται με την πολιτική αλλά και με τα οικονομικά λένε αποδοτικότητα ίσον ενεργειακή αποδοτικότητα. Βεβαίω, είναι σημαντικό τμήμα τη. Αλλά όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι η αποδοτικότητα των πόρων είναι πολύ ευρύτερο θέμα. Για παράδειγμα, η διαχείριση των υδάτων, των εδαφών, των ωκεανών. Όλα αυτά επίση παίζουν μεγάλο ρόλο. Και ελπίζω αυτή η αποδοτικότητα των πόρων, η μεταβατική πλατφόρμα για την αποδοτικότητα των πόρων και η δημοσιότητα που θα δώσουμε σε αυτήν θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε την πολιτική αποφασιστικότητα για το θέμα αυτό. Αναφερθήκατε επίσης σε κάτι που μου φαίνεται πολύ ελκυστικό που θα μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε και σε αυτή την πλατφόρμα για την αποδοτικότητα. Αν μπορούμε να εφαρμόσουμε δηλαδή μια ιδέα που θα βοηθούσε σε καλύτερες πρακτικές εφαρμογής. Πολλοί ελκυστική, πολύ λογική. Έχει έννοια. Ε, τα υπολείμματα φαρμακευτικών στα ύδατα που αναφέρθηκαν διάφοροι συνάδελφοι, ο κ. Ρώση και εσείς, Βεβαίως, το πρότυπο που έχουμε υπόψη μας δεν αντιμετωπίζει συγκεκριμένα αυτό, αλλά όπως ξέρετε πρόσφατα κάναμε μια πρόταση για να ενημερωθεί ο κατάλογος χημικών ουσιών στα ύδατα και για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνονται τρεις φαρμακευτικές ουσίες που έχουμε συγκεκριμένες ε, πληροφορίες ότι είναι επικίνδυνες. Είναι ένα νέο βήμα. Βεβαίως θα γίνει σοβαρή συζήτηση για το θέμα αυτό, αλλά ελπίζω ότι θα περάσει. Η ενημέρωση πρέπει οπωσδήποτε να γίνει στα πλαίσια της οδηγίας ε, πλαίσιο για τα ύδατα. Συνδυάζεται λοιπόν με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας, διότι δεν έχει προχωρήσει και τόσο πολύ η εφαρμογή, πρέπει να το πω ειλικρινά. Η μόλυνση μέσω χημικών ουσιών των υδάτων πρέπει να είναι στο κέντρο της προσοχής μας, σας διαβεβαιώ ότι θα είναι. Η τελευταία ερώτηση, Ματία, ήταν για τη φορολογική πολιτική. Αυτό είναι ίσως πιο εύκολο κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσω αυτής της διαδικασίας εξαμήνων δεν θα πρέπει να πω πολλά γιατί δεν ξέρω ακριβώς τι θα είναι στην ε, πρόταση που θα κάνουμε αύριο αλλά το συζητήσαμε και κάποιες συστάσεις οπωσδήποτε θα προτείνουν τα κράτη-μέλη να περάσουν από τη φορολόγηση της εργασίας στη φορολόγηση στην περιβαλλοντική φορολόγηση. Δεν θέλουμε να αυξηθεί ο όγκος της φορολόγησης. Αυτό είναι σίγουρο. Εάν κάτι ισχύει στην Ευρώπη είναι σίγουρα ότι η τιμή της εργασίας, το εργατικό κόστος είναι υψηλό. Και δεν θέλουμε να αυξηθεί. Θέλουμε λοιπόν να μεταφέρουμε τη φορολόγηση. Αλλά αν ε, κάποια κράτη-μέλη χρειάζονται συμπληρωματικού πόρους, που νομίζω ότι όλα τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή χρειάζονται συμπληρωματικού πόρους, Καλύτερα λοιπόν θα ήταν οι φόροι να αφορούν την περιβαλλοντική εφαρμογή και όχι το εργατικό κόστος. Και οι επιδοτήσεις για το περιβάλλον είναι φοραβαλλαγές πολλές φορές. Είναι λογικό. Ξέρετε πόσο κρίσιμη είναι η περίοδος για την οικονομία μας. Έχει λοιπόν έννοια να αντιμετωπίζονται προβλήματα έτσι. Γιατί έτσι, χωρίς να αυξάνουμε τη φορολογία, βελτιώνουμε το περιβάλλον. Η εσωτερικοποίηση του κόστους βεβαίως είναι η σωστή λύση. Βεβαίως, ε, οι καταναλωτές αντιδρούν στα κίνητρα που τους δίδονται μέσω των τιμών οπωσδήποτε πρέπει να ε, οδεύσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δεύτερος γύρος ομιλητών. Αλλά πρώτα να καλωσορίσω ένα νέο συνάδελφο από την Πορτογαλία, Άλτα Σούζα. Νέος αναπληρωματικός, καλώς ήρθατε. Νέα αναπληρωματική. Δεύτερος γύρος ερωτήσεων. Πρώτος ομιλητής, Χαρχάινς Φλόρεντς. Α, έχετε δίκιο. Πρώτα ο Επίτροπος να κάνει μια εισαγωγή. Για το Ρίο. Τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για τη συνεισφορά του όσον αφορά την τοποθέτησή μας ενώπιση του 2020 είχαμε γερή διαπραγματευτική θέση. Ξέρω ότι δεν θέλατε επίσημα να παρουσιαστούν στη διάσκεψη θέση σα, αλλά αν μη τι άλλο φροντίζω να ενημερώνεστε σωστά και όσοι από εσά ε, είσαστε εκεί και με του οποίου συναντηθήκαμε ε, την προηγούμενη εβδομάδα θα το θεωρήσουν κάτι πολύ θετικό. Μπορείτε να βασιστείτε σε εμά. Με όποιο τρόπο και αν ε, εκπροσωπηθείτε, μπορείτε να βασιστείτε σε εμά. Το θέμα των δαπανών. Εμεί θα χρησιμοποιήσουμε τη συμμετοχή μα όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις και τις ε, δραστηριότητες κατά προτεραιότητα βάσει της ανακοίνωσής μας. Το Κοινοβούλιο ζήτησε οι διασκέψεις Ρίο Συνήκωση να καταλήξουν σε αυτά αποτελέσματα, να πετύχουν τους στόχους ε, και να τεθούν νέοι πολύ συγκεκριμένοι. Κύρια προτεραιότητά μας λοιπόν για το είναι να συμφωνήσουμε για συγκεκριμένε δράσει και στόχου. Οι προτάσει μα έχουν να κάνουν με την αηφόρα ανάπτυξη, με οικοσυστήματα για τους ωκεανού και τα απόβλητα και όλα αυτά τα θέματα αναφέρονται και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι προτάσει αυτέ είναι πολύ βασικές για να καταπολεμήσουμε την ένδια, για να ενισχύσουμε την πράσινη οικονομία και να προσφέρουμε ευημερία με νέες θέσεις απασχόλησης, ενίσχυση της κοινωνικής ε, διάστασης. Θέλουμε πράσινη οικονομία για όλους και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τρόπο στεναρό διάφορε συνήθειε που έχουμε μέχρι τώρα και πρέπει να δούμε πώς θα πετύχουμε την αηφόρο ανάπτυξη παντού. Προστασία της γης, των οικοσυστημάτων, του εδάφους δηλαδή, είναι κάτι πολύ βασικό αν θέλουμε να έχουμε και διατροφική ασφάλεια και να καταπολεμήσουμε την ένδια. Όλα αυτά εξαρτώνται από τα οικοσυστήματα. Αν ε, μπορούμε να έχουμε έναν σημαντικό ρόλο για το πρασίνισμα της οικονομίας, αυτό είναι πολύ σημαντικό και για να προωθήσουμε τους στόχους μας στο Ρίο. Το Ρίο, στο Ρίο επίσης θα υπάρξουν και οι ε, αεφόροι στόχοι. Οι δικοί μας στόχοι για την πράσινη οικονομία πιστεύουμε ότι μπορούν πολύ καλά να συμπεριληφθούν στην όλη διαδικασία. Θα, ενισχύσει, θα ενισχύσουμε λοιπόν και τους στόχους της χιλιετίας και θα φροντίσουμε και για την περίοδο μετά του 2050 ενισχύοντας την αηφόρα ανέπτυξη και συμπληρώνοντας την με συνολικό τρόπο για τι συστάσεις. Πρέπει να κινητοποιήσουμε όλου του πόρου που έχουμε σε εθνικό, διεθνέ επίπεδο, ιδιωτικού δημόσιου, και θα συνεχίσουμε να ε, προχωρούμε προ του συμφωνημένους στόχου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίση συμφωνεί με τη δημιουργία μια υπηρεσία για το περιβάλλον όπως έχει πει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στηρίζουμε και ευρύτερε μεταρρυθμίσεις για το ε, θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά την αηφόρα ανάπτυξη. Αυτό που μου απασχολεί είναι ο αργός ρυθμός διαπραγματεύσεων. Κάτι το οποίο μας δυσκολεύει να πετύχουμε τους στόχους μας. Μετά το Ρίο, μην ξεχνάμε ότι το μήνυμα του Κοινοβουλίου αυτού ήταν η αηφόρος ανάπτυξη που θέλετε να μπει στην πρώτη γραμμή σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλουμε λοιπόν να είναι συνεπής η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να έχει κάποιο νόημα το αποτέλεσμα του Ρίο. Και βασιζόμαστε στη δική σας στήριξη και γι' αυτό. Δύο λόγια τώρα για το είδωρ. Θα δημοσιευθεί τον Νοέμβριο κάτι σχετικό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε ε, παρκείς ε, και αποδοτικούς πόρους ύδατος. Και για να το πετύχουμε θέλουμε διαδραστικές ε, ενέργειες και συμπλήρωση του τωρινού πλαισίου. Όσον αφορά τώρα την τρίτη διάσκεψη για το είδωρ, και εδώ θα συζητηθούν οι διάφορες επιλογές με τους εταίρους μας. Αλλά έχουμε και διαβούλευση η οποία τρέχει και θα κλείσει σύντομα. Είναι πολύ βασικό και αυτό για το blueprint, για το πρότυπο. Πιστεύω θα έχετε δει και εσείς την έκθεση του κυρίου Σίμπερ. Περιμένω και τις δικές σας απόψεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να δώσουμε σάρκα και οστά στις προτάσεις μας. Έχουμε εγκρίνει ε, και άλλα πράγματα για το είδωρ. Χρειαζόμαστε καινοτόμε λύσει. για να αντιμετωπίσουμε τις διάφορε προκλήσεις που έχουν να κάνουν με το είδωρ. Και έπειτα υπάρχουν και οι αγορέ σχετικά με την καινοτομία για το είδωρ, κάτι το οποίο χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και με ιδέες που μας έρχονται από αλλού. Τη Δευτέρα ήμουνα στην Δανία και είδα και εκεί τι αντλίες ύδατος φτιάχνουν και τι αποτελέσματα έχουν. Το θέμα της αποδοτικότητας του ύδατος και της ποιότητας του ύδατος είναι κάτι που μας ενδιαφέρει γενικότερα. Υπάρχουν λοιπόν και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και από εδώ και πέρα περιμένω τις δικές σας απόψεις για όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Dank. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα Ρίο συνήκωση Αυτό καθε αυτό, αλλά και η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου θα πρέπει να το συζητήσουμε και σε άλλα επίπεδα, δηλαδή Κοινοβούλιο και Επιτροπή. Νομίζω ότι και ο κύριος Σεύκοβιτς είναι ο κύριος συνομιλητής για το πώς θα μπορέσει να συμμετάσχει πλήρως στο Κοινοβούλιο, να εντάσσεται πλήρως στο Κοινοβούλιο σε αντιπροσωπείες της Κομισιόν και του Συμβουλίου για να μπορεί επιτόπου να εργάζεται σωστά. Γιατί σε τελευταία ανάλυση, αν πρέπει να παίρνει αποφάσεις η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου που θα πρέπει να τις ε, υπερασπιζόμεθα ενώπιον των εκλογέων μας, τότε πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Με τι τρόπο μπορεί σωστά να συμμετέχει σε αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Κοινοβούλιο, να μπορεί επιτόπου δηλαδή να εργάζεται σωστά και όχι να υπάρχουν τρία-τέσσερα τμήματα της αντιπροσωπείας της Ένωσης. Οπότε, ο κύριος Ζέμπερ. Μία ερώτηση. Κύριε Επίτροπε, υπάρχουν φήμες ότι η Κομισιόν έχει κλείσει για το Ρίο 120 δωμάτια. 120. Ισχύουν αυτές οι φήμες ή είναι μόνο φήμες. Θα με ενδιέφερε. Γιατί εμείς ως Επιτροπή δεν πηγαίνουμε. Νομίζω ότι θα έπρεπε να διευκρινιστεί αυτό. Λοιπόν, αν ήξερα τι κάνουν όλοι και όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία θα ήμουν μάγος. Είπα ότι εδόθη ένα σωστό μήνυμα από το Κοινοβούλιο και επομένως το σαφές μήνυμα που στείλαμε προς τις υπηρεσίες μας και τις άλλες υπηρεσίες ήταν ότι θα πρέπει να ενεργήσουν αναλόγως και με τρόπο υπεύθυνο σχετικά και με την ε, ιδιαίτερη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο. Πρέπει να σας πω πάντως ότι θέλουμε να πάμε στο Ρίο, ε, θέλουμε να έχουμε μαζί μας το Ρίο όσους μπορούν να μας βοηθήσουν έτσι ώστε να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Πρώτος ομιλητής, ο Ζάλφος Καλχάινς Λόρεντς. Κύριε Επίτροπε, έχω ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα. Είστε ο αγαπημένος μου επίτροπο. επίτροπος. Αλλά έχω ένα πρόβλημα με την γενική σας διεύθυνση. Δεν μ' αρέσει η ανακοίνωση ότι επίκυνται τόσα νέα νομοθετήματα. Βεβαίως όλα αυτά είναι αναγκαία. Αλλά αν ρεαλιστικά δω τι έχουμε εφαρμόσει, τότε αυτό είναι κόλαφος. Κάθε φορά τόσα θέματα. Για παράδειγμα, η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα είναι καταστροφή. Όλοι μπορούμε να συγχαίρουμε ένα τον άλλον. Αλλά να πάμε σε κάποιο σύνορο, εκεί που ο ε, Μοζέλας περνάει από μια χώρα στην άλλη ή ο Ρήνος. Να δείτε τι τιμές υπάρχουν μέσα στα νερά αυτά που απαγορεύονται στη χώρα όπου μπαίνει το ποτάμι. Και η Κομισιόν δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί είναι τόσο ευρέως ορισμένες οι έννοιες που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Έχετε λοιπόν καθήκοντα ελέγχου ως Επιτροπή. Πρέπει να αλλάξετε κάποιες οδηγίες. Γιατί όπως είναι τώρα οι οδηγίες μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Η Ιταλία κάνει ό,τι θέλει. Ε, ορίζουν ούτω τα απόβλητα και η Επιτροπή μπορεί να έρθει και της λένε κοιτάξτε είναι εθνικό καθήκον να ορίσουμε τι είναι απόβλητα. Ο Κρις Ντέιβις μίλησε για τα αυτοκίνητα. Η κατάσταση είναι όντως άθλια. Γιατί σε τελευταία ανάλυση ο κάθε οδηγός μπορεί να καθορίσει αν το αυτοκίνητό του μπορεί να βγει στον δρόμο ακόμη και αν δεν έχει λάστιχα. Η κατάσταση λοιπόν είναι απελπιστική. Όλη η κατάσταση με τα οχήματα, με τα οχήματα που είναι παλιοσίδρα στην ουσία, πηγαίνουν στην Ανατολική Ευρώπη και υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προσαρμοστεί για ε, έχουν, οι εταιρείε που έχουν προσαρμοστεί για την ανακύκλωση των υλικών τους χρεοκοπούν διότι δεν παίρνουν παλιά αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα αυτά εξακολουθούν να κυκλοφορούν. Έχουν γίνει πολύ άσχημα πράγματα. Και κοιτάξτε, η επιθυμία μου είναι. Μιλάμε όλοι για, την, για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά είναι γελία η κατάσταση. Κοιτάξτε όμω, ο τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται αυτό είναι εντελώ διαφορετικό στην Ολλανδία από ό,τι είναι στη Γερμανία. Σα παρακαλώ, να κάνουμε λιγότερα, να τα κάνουμε καλύτερα γιατί έτσι θα μας καταλαβαίνουν και καλύτερα οι πολίτες. Είμαι λοιπόν σε μια αντιφατική κατάσταση. Αλλά ενώ ε, χαίρομαι για τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε, ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζει η Κομισιόν τις αρμοδιότητες του δεν είναι καλή. Ευχαριστώ. Μέρκης. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας συγχαρώ διότι αγαπητοί συνάδελφοι, όχι μονάχα σήμερα στην δική μας Επιτροπή μπορείτε να θέσετε ερωτήματα στον Επίτροπο, αλλά απαντάει, δέχεται και απαντάει ερωτήματα στο Twitter. Ε, εγώ υπέβαλα δύο ερωτήσεις την Παρασκευή και μου απέντησε αμέσως. Συγχαρητήρια λοιπόν και γι' αυτό. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν κάποια ε, ζητήματα τα οποία ε, φαίνονται μικρά αλλά μπορεί να έχουν πάρα πολύ μεγάλο ε, αντίκτυπο. Η βιομάζα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα και στην έκθεση και μπράντε. Πότε θα σταματήσει η αποτέφρωση των ανακυκλώσιμων υλικών που σε πολλές περιπτώσεις μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν ε, για άλλους σκοπούς. Ε, η απαγόρευση των χωματερών που έχει ζητηθεί ήδη επανειλημμένα και το ζητάμε και στην έκθεση Γεμπράντε, τελικά θα έχει ο τέλος στην νομοθεσία μέχρι το 2020. Επίσης, ε, λέτε ότι ε, ε, η απομάκρυνση των φαρμακευτικών ε, ουσιών λέτε ότι είναι μόλυνση, όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως κάποιες φορές αυτά, αυτές οι ουσίες, αυτά τα υλικά. Επομένως, εάν, εάν ε, ε, θεωρηθούν απόβλητα και αποβληθούν άμεσα από τις νοσοκομιακές μονάδες, ας πούμε, ενδεχομένως θα χάσουμε ε, κάποιες ουσίες. Και βεβαίως το ίδιο ισχύει, με προβληματίζει επίσης η περιεκτικότητα σε φωσφορούς ουσίες και σε αντιβιωτικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μπουκαλάκι με το αγαπημένο σας, με την αγαπημένη σας ουσία, το νερό. Γιατί λοιπόν αυτά τα κουβαλάμε, τα νερά και τα μπουκαλάκια από το ένα μέρος της Ευρώπης στο άλλο, ενώ στην ουσία ε, είναι περίπου καθαρό νερό της βρύσης, οποίο, με το οποίο γεμίζονται, γιατί τα συστατικά είναι περίπου όμοια. Ε, γιατί λοιπόν τα κουβαλάμε δημιουργώντας ε, τέτοιο, τόση μόλυνση με διοξίδιο του άνθρακος. νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι και έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες προσπάθειες έτσι ώστε να μην επιτρέπονται πλέον αυτά τα μπουκαλάκια. Κάντε κάτι και γι' αυτό λοιπόν λοιπόν. Επίσης, ε, η διάλυση των ε, νανοστοιχείων Μία ερωτησούλα ακόμα μόνο, γιατί φτάνουμε τώρα σε αυτά τα μικρά στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχουν ε, λοιπόν ε, στοιχεία που έχουν βρεθεί αργύρου και τα λοιπά που μπορεί να είναι ε, πολύ επικίνδυνα. Δεν είναι βέβαια σε όλα τα είδη μπουκαλιών, σε ορισμένα, αλλά παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Αυτά τα στοιχεία θα ληφθούν υπόψη και στις νομοθετικές προτάσεις και να μην μείνουν μονάχα στη στρατηγική. Ευχαριστώ που τηρήσατε για τα δύο λεπτά. Αλλά κοιτάξτε, εδώ αυτό που έγραψε ο Επίτροπος στο Twitter είναι υποδηματικό εγώ και εγώ παρακολουθώ τα tweet ε, του κυρίου Ποτότσνικ. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να εκφραστεί μέσω των ε, κοινωνικών ε, μέσων. Είναι πολύ καλός τρόπος, υποδειγματικός, να έρχεται σε επαφή με τους πολίτες. Και Μπράντι, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που ήρθατε και ευχαριστώ και για την συνεργασία σας με την άτυπη αυτή η αντιπροσωπεία στο Ριό. Χαίρομαι που θέλετε να συνεργαστούμε στενά μεταξύ μας. Προσωπικά πιστεύω ακόμα ότι δεν είναι πολύ αργά αυτή η άτυπη αντιπροσωπεία με κάποιο τρόπο να γίνει μια επίσημη αντιπροσωπεία, αλλά αυτό είναι μάλλον μια άλλη συζήτηση. Σήμερα ακούσαμε ότι στη Γερμανία ε, πέτυχαν ένα παγκόσμιο ρεκόρ όσον αφορά την ε, ενέργεια που παράχθηκε από, την, από τον ήλιο, χάρη στον καλό καιρό. 22.000 ΜΒ αν δεν απατώμε. Κάτι το οποίο αντιστοιχεί σε 20 πυρηνικούς σταθμούς. Απίστευτο, ε! 50% της συνολικής κατανάλωσης ενέργεια παρήχθη από τη ηλίκη αυτό το Σαββατοκύριακο. Και εγώ με το Twitter πήρα απάντηση από κάποιον, όπως είπε ναι, αλλά με τι κόστος. Είναι ένα παράδειγμα όμως, τόσο όμορφο παράδειγμα μιας καλής ιστορίας για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και έχετε τέτοια ανταπόκριση για μένα είναι πολύ βασικό οι χώρες μέλη να μπορέσουν να αντιδράσουν αποτελεσματικά. Έχω την αίσθηση ότι η γενική εντύπωση για το πόσο επήγει το θέμα και το θετικό πνεύμα ε, που θα έπρεπε να υπάρχει δεν είναι ακόμα παρόν. Ίσως εσείς μπορείτε να βοηθήσετε επηρεάζοντας τα κράτη-μέλη εν ώψη του ριού. Τώρα που μιλάμε, τι γίνεται στη Νέα Υόρκη που έχουμε τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων. Τέλος, οι RG, οι χώρες που θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας στο Ρίο. Μήπως θα γινόταν αν μετά το Ρίο, ακόμα και αν δεν πετύχει το Ρίο, να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα συνασπισμό εκείνων των χωρών που θέλουν να προχωρήσουμε με την αηφόρα ανάπτυξη έτσι όπως εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει. Και μήπως θα μπορούσαμε ε, να δίναμε κάποια εμπορικά πλονεκτήματα με αυτόν τον συνασπισμό ε, χωρών που θέλουν κίνητρα ώστε να προχωρήσουμε σε αυτά που θέλουμε και που πιστεύουμε ότι γι' αυτά οργανώνεται και η διάσκεψη του Ρίο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κατρίν από τους πράσινους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε για το briefing και ευχαριστούμε και για αυτές τις πιστοποιήσεις ε, οι οποίες ε, θα μας ε, δώσουν την δυνατότητα να παραστούμε σε τις συναντήσεις του Ρίο με ανεπίσημο τρόπο και θα μπορείτε να βασίζετε πάνω μας οπωσδήποτε για οποιαδήποτε βοήθεια και άλλωστε είπατε ότι η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπνέεται τα μάλα από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είχα μια ερώτηση όσον αφορά την προετοιμασία της διασκέψεως κορυφής, γιατί υπάρχουν αρκετά στοιχεία τα οποία θεωρώ ανησυχητικά. Μεταξύ αυτών ε, πρώτο είναι το εξής. Διάβασα δυστυχώς στο γαλλικό τύπο μία δήλωση της βραζιλιάνικης κυβέρνησης ε, που ε, ανακοίνωσε ότι οι στόχοι του 2012 δεν θα είναι τόσο περιβαλλοντικοί, θα είναι κυρίως οικονομική σε αντίθεση με το πρώτο ρίο. Επομένως προκύπτει το πρώτο ερώτημα. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμείς έχουμε επανειλημμένα προσπαθήσει να δούμε τι σημαίνει πράσινη οικονομία και τι πρέπει μπορεί να καλύπτει, άρα αυτό θα συζητηθεί. Όμως, πού βρισκόμαστε σήμερα ε, στις διαπραγματεύσεις, έχουμε προχωρήσει, αυτή η πράσινη οικονομία είναι όντως αυτή η πράσινη οικονομία την οποία έχει στο νου του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, που θα βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, ε, που θα λαμβάνει υπόψη και την διατήρηση των πηγών αλλά και την, το καλό της κοινωνίας. Μετά την πρώτη διάσκεψη για τη γη στην νομίζω ότι δεν έχουν ακόμα λυθεί τα βασικά οικολογικά ζητήματα και δεν μπορούμε ακόμα με συγκεκριμένο τρόπο να συνδέσουμε την οικονομική κρίση με, την, το πρασίνισμα της οικονομίας. Δεν έχουμε ακόμα πείσει ότι θα πρέπει να αλλάξει, ε, ότι μπορεί να, να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση μέσα από τροποποίηση του μοντέλου. Ε, επίσης, ε, φαντάζομαι ότι θα γίνει λόγος ε, για το θέμα της ε, καταστροφής των δασών στην Βραζιλία. Έχουμε έναν νέο ε, δασικό νόμο ε, που μας απασχολεί πάρα πολύ και μας ανησυχεί. Για να επανέλθω στην πράσινη οικονομία, να πω ότι στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαμε αναφερθεί στην, σε τα στοιχεία κοινής ωφελίας τι κάνουμε λοιπόν όσον αφορά π.χ. το καθεστώς των περιβαλλοντικών προσφύγων, όσον αφορά την μη δυνατότητα τεχνίας για ορισμένες ανακαλύψεις. Τι έχουμε κάνει για όλα αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ γιατί δεν ξεπεράσατε τα δύο λεπτά. Ε, γύρω ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ ε, να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την ε, παρουσία του ε, και για τα όσα μας είπε ενημερωτικά. Δεν συμφωνώ απολύτως με τον Σάνχο Γιομπράντι όταν μιλάει για την ηλιακή ενέργεια ε, γιατί ξέρω ότι δημιουργούνται και προβλήματα ε, και δημιουργούνται και προβλήματα στις ε, εταιρείε που ασχολούνται με την ενέργεια στην χώρα μου και επομένως μπορούν να δημιουργηθούν πολλές ανισορροπίες στην Ευρώπη. Θα ήθελα εγώ να μιλήσω για το Ρίο συν 20. Το Κοινοβούλιο δεν, ε, δεν θα έχει την δυνατότητα να εκφραστεί σαν αντιπροσωπεία ε, στο Ρίο και ε, Χαίρομαι που αναφέρατε το ενδεχόμενο συμμετοχής μας ως μη επίσημης αντιπροσωπείας. Ανεξάρτητα από το αν είμαστε παρόντες φυσικά ή όχι, οπωσδήποτε ε, ε, θα πρέπει εκ των υστέρων να έχουμε πλήρη ενημέρωση και να ενημερώσουμε και παραέξω για τα όσα θα έχουν λάβει χώρα στη διάσκεψη του Ρίο. Μία ερώτηση ήθελα να κάνω για το νερό το θέμα των υδάτινων πόρων, γιατί το πρόβλημα αυτό είναι κατεπήγον στην Ευρώπη, αλλά ακόμα πιο επίγον στις αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως όσον αφορά το πόσιμο ύδρο. Λέμε ότι σαν αναπτυγμένη και πλούσια Ευρώπη θα πρέπει να βοηθάμε την λιγότερο, τον λιγότερο αναπτυγμένο και φτωχό ε, νότο. Πιστεύετε ότι για μία ακόμα φορά θα έχουμε κάποιες γενικές δηλώσεις για την στήριξη προς αυτές τις χώρες ή θα μιλήσουμε πλέον για συγκεκριμένη τεχνολογική υποστήριξη για το πόσιμο είδωρο. Άνθος Κόκοβιτς. Κύριε Επιτροπέ, Είμαι σε μια ιδιαίτερα δυσχερή κατάσταση. Στη ζωή χρειάζεται εργασία, δημιουργικότητα και υγεία. Πώς μπορούμε να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα στοιχεία. Την υγεία μας ε, τη σκεφτόμαστε μόνο όταν τη χάσουμε. Στην οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε στην παρούσα φάση. Ε, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε αλλά ε, θα πρέπει και η οικονομία μας και οι επιχειρήσεις μας να μπορούν να επιβιώνουν. Επειδή λοιπόν υπάρχει κρίση, βεβαίως πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε την αηφορία. Αλλά παράλληλα να είμαστε και ρεαλιστές. Γιατί η Ευρώπη βεβαίως ε, είναι προτεργάτη στη χρήση περιβαλλοντικής τεχνολογίας και βεβαίως ε, το επιτυγχάνουμε θαυμάσια, αλλά αυτό μπορεί να μας δώσει ευκαιρίες και στην οικονομία. Είναι ενδεχομένως ένας τομέας όπου μπορούν επιτυχώς να δράσουν οι επιχειρήσεις μας. Αλλά βεβαίως όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να φέρουν το κόστος ε, της χρήσης των αποβλήτων τους, των υδάτων για παράδειγμα. Πρέπει να γίνει ένας επανυπολογισμός. Να δούμε τι εξακολουθεί να είναι ρεαλιστικό. Στη χώρα μου, στη Σλοβενία ξέρετε, Έχουμε πολύ νερό. Έχουμε πολλούς φυσικούς πόρους. Και μπορούμε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε το, τα ύδατά μας και για την παραγωγή ηλεκτρικού, αλλά και στον τουρισμό φυσικά, σε πολλούς τομείς ε, χρησιμοποιούμε τους υδάτινους πόρους μας. Εν ώψη του ορίου, πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει περισσότερη ισορροπία Βεβαίως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, αλλά εκτός από την οικονομία πρέπει να ε, ε, φροντίσουμε και το περιβάλλον. Ευχαριστώ, Σανώνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε για τα ενδιαφέροντα εισαγωγικά που μας είπατε. Με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον παρακολούθησα ε, την πρόθεση την οποία ανακοινώσατε εσείς ε, να ανακοινωθούν νομοθετικές προτάσεις ε, που εξαιρετικά ενδιαφέροντες με βέβαιος μέχρι το τέλος του 2013 από την Κομισιόν. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο κατέδειξαν και άλλοι συνάδελφοι, το θέμα της εφαρμογής, της υλοποίησης των οδηγιών. Αναφέρομαι κυρίως στην οδηγία για το νερό ε, για την οποία πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα ε, δεν την έχουν ακόμα ενσωματώσει, δεν, την έχουν, δεν έχουν ακόμα κάνει ταυτοποίηση το, του υδροφόρου ορίζοντα και των ε, λεκανών απορροής, δεν έχουν δώσει συγκεκριμένο πρόγραμμα εκμετάλλευσης των υδάτινων πόρων και επίσης δεν έχουν υποβάλει πρόγραμμα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, για την εξυγίανση ε, του υδροφόρου ορίζοντα. Ε, ειδικά στην περιοχή από την οποία προέρχομαι εγώ, δηλαδή η ε, παιδιάδα του Πάδου, έχει εξαιρετικά βεβαρημένο υδροφόρο ορίζοντα. Η το υπέδαφος έχει μολυνθεί, τα ύδατα τα υπόγεια έχουν μολυνθεί και κανένας δεν προσπαθεί ε, να τα εξηγιάνει ή δεν προτίθεται από ό,τι φαίνεται και όλα αυτά πιστεύω ότι είναι επίπτωση και απόρρια της ε, μη εφαρμογής της οδηγίας. Θα πρέπει η Κομισιόν με κάποιο τρόπο να ασκήσει πίεση. Με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον ακούω όλα αυτά που λέτε για το blueprint, για το νερό κτλ. Αλλά εάν ζητήσει το Κοινοβούλιο κάτι από τα κράτη-μέλη και εξακολουθεί να κάνουν τον κουφό κάποια ε, κράτη-μέλη. Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Θα είναι ότι θα δημιουργηθεί μεγάλη ανισορροπία και ανισότητα μεταξύ χωρών, μεταξύ πολιτών εν τέλει. Γιατί ε, θα ε, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα έχουν ένα καλό ε, υδροφορορίζοντα και αυτοί οι οποίοι θα εξακολουθούν να έχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα όσον αφορά τον έλεγχο των υδάτων. Επομένως κάτι πρέπει να γίνει όσον αφορά την εποπτεία, τον έλεγχο και τις κυρώσεις Επίση, ενδεχομένως. Επίσης, προηγουμένως αναφερθήκατε και στην οδηγία για, τον, για την ποιότητα του αέρα και τον ατμοσφαιρικό αέρα. Και εδώ όμως, στην προκείμενη περίπτωση, υπάρχουν ε, περιοχές ε, της Ευρώπης ε, στις οποίες οι πολίτες αναπνέουν μολυσμένο δηλητηριώδη αέρα. Έχουμε την ε, έκθεση Γκεμπράντι, ε, την οποία εγκρίναμε ε, πριν από μερικές μέρες. Ας ξεκινήσουμε από εκεί λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε επίσης από το να σταματήσουμε πλέον μία και καλή την αποτέφρωση. Πώς είναι δυνατόν να συνεχίζουμε την αποτέφρωση η οποία ξέρουμε ότι εκλεί, προκαλεί μάλλον την έκκληση τόσων αερίων τη στιγμή που κάνουμε τόση συζήτηση για μία Ευρώπη ελεύθερη από διοξίδιο του άνθρακα. Αυτά περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Για να απαντήσει ο κύριος Επίτροπος, παρακαλώ. Πολλής λόγος έγινε για την υλοποίηση. Πολλά υπόθηκαν όσον αφορά την εφαρμογή. Συμφωνώ με τα τελευταία σας συμπεράσματα που ήταν ε, ότι οι αλλαγέ είναι αναγκαίες. Συμφωνώ. Συμφωνώ ότι όντω πρέπει να προχωρήσουμε στι ε, αλλαγέ που θα κάνουν τη δράση μα πιο αποτελεσματική. Όσον αφορά τώρα τη διαχείριση και την υλοποίηση τη οδηγία για το ύδατα. Ένα από τα θέματα είναι το πρότυπο πάνω στο οποίο δουλεύουμε. Αναλύουμε ε, ενδελεχώς όλες τις προτάσεις, μία προς μία. Και θα δώσουμε την τελική μας απάντηση, τι πρέπει να γίνει. Ο λόγος είναι ότι ξέρουμε ότι είμαστε στη φάση της υλοποίησης, η οποία όμως ακόμα δεν μας δημιουργεί αρκετή εμπιστοσύνη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της οδηγίας αυτής. Για να γίνω όμως κάπως πιο ειδικό. Όπως είπατε σωστά, δεν έχουμε τη δυνατότητα τώρα να πάμε και να δούμε, μετρήσουμε τι υπάρχει μέσα στο νερό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι κάτι που κάνουν τα κράτη-μέλη. Και στην ομοθεσία αναφέρεται ξεκάθαρα και με ποιο τρόπο πρέπει να μας μεταφέρουν τα αποτελέσματα. Περιμένουμε έτσι καλώς όσον αφορά την ε, ρήπανση του αέρα, τα αποτελέσματα τα περσινά. Και κάθε φορά 10 μήνες αργότερα παίρνουμε τα αποτελέσματα από τις εκάστοτε μετρήσεις. Συνεπώς, όλα αυτά είναι κάπως μακριά από την ε, πραγματική κατάσταση ως έχει. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που θα ήθελα να αντιμετωπίσω. για την βιομάζα. Εξήγησα ήδη. Για την απαγόρευση. Κάτι σημαντικό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι στο χάρτη πορεία λέει ότι 2020 θα έχει πάψει οι χωματερέ για τα υλικά αυτά κτλ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει να αναθεωρήσει την επαναχρησιμοποίηση ε, και τους διάφορους ε, στόχους οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ανακύκλωση και με τα απόβλητα για να φτάσουμε σε μηδενικές τιμές έτσι όπως προβλέπετε. Οπότε ναι, δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Αυτός ε, είναι ο στόχος. Για τα πλαστικά και για όλα τα ειδικά θέματα τα οποία ανέφερες. Ο κανόνας που ακολουθούμε στις νομοθετικές μας προτάσεις είναι να υπάρχουν αρκετές επιστημονικές αποδείξεις, να έχουμε αρκετά στοιχεία και να μπορούμε να βασιστούμε στο ότι αυτό που προτείνουμε θα λειτουργήσει. Μερικές φορές όταν δεν γίνεται αυτό, πιέζουμε περισσότερο για μελέτες ή κάνουμε περισσότερα πράγματα. Έτσι κι πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα προτείνουμε κάτι λάθος. Για τα πλαστικά μπουκάλια, το μόνο που έχω να πω είναι ότι ότι η νομοθεσία είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να φροντίσουμε να τίθεται και σε εφαρμογή. Υπάρχει η νομοθεσία για την εσωτερική αγορά, για παράδειγμα. Είναι πράγματα αυτά τα οποία αποτελούν την πραγματικότητά μας. Και ξέρετε ότι η εσωτερική αγορά είναι αυτή που είναι. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε την ε, μεταφορά τέτοιων μπουκαλιών η παραγωγή που παράγουν στο Βέλιο θα έπρεπε να προσφέρουν τις καλύτερες τιμές, άρα και αυτούς να προτιμάμε. Γιατί έχουν χαμηλότερο κόστος να μεταφέρουν εδώ τα μπουκάλια. Πας περιπτώσει τις ανησυχίες σου πάντως τις σέβομαι απόλυτα και τις σημειώνω. Τώρα, για την ηλιακή ενέργεια. Αν με ρωτήσετε, εγώ έτσι καλώς είμαι υπέρ της έρευνας, θα βάζα στοίχημα, αν και δεν θα ζήσω για να δω το αποτέλεσμα, ότι σύντομα η ενέργεια που θα χρησιμοποιούμε θα είναι ηλιακή. Αυτά είναι μαθήματα που παίρνουμε από τη φύση. Η φύση μας διδάσκει. Και ίσως αυτό είναι που δεν κάνουμε αρκετά, δεν σκεφτόμαστε αρκετά, δεν κοιτάμε αρκετά τη φύση για να πάρουμε μαθήματα από αυτήν. Εγώ βάζω στοίχημα, αλλά δυστυχώς δεν θα είμαι εδώ για να δω και το αποτέλεσμα. Τώρα, τι ρόλο παίζουν τα κράτη-μέλη στο ΡΙΟ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο ισχυρή όσοι είμαστε ενωμένοι. Όλοι θα μπορέσουν να δουλέψουν, όλες οι χώρες έχουν δουλειά να κάνουν και είναι ζωτική σημασία να μεταφέρουμε το ίδιο μήνυμα εκεί μια ισχυρή Ευρώπη δεν θα αγνοηθεί και θα οδηγήσει σε αλλαγές. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όσον αφορά την Νέα Υόρκη, σήμερα ξεκίνησαν τη συζήτηση. Οπότε σήμερα το βράδυ θα ενημερωθώ, άρα δεν μπορώ εγώ να σας ενημερώσω. Δεν γνωρίζω τι έχει γίνει. Ξέρω ότι υπάρχει ένα νέο σχέδιο στο τραπέζι από τον πρόεδρο Και η πρώτη εκτίμηση λέει ότι πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Για τον συνασπισμό τώρα στον οποίο αναφερθήκατε χωρών που θέλουν να προχωρήσουν. Εντάξει, πάλι θα σας απαντήσω, ας πετύχουμε στο Ρίο. Αν κατά σύμπτωση δεν το πετύχουμε αυτό, τότε βλέπουμε για τα παρετέρω. Το πρόβλημα το οποίο αναφέρεται η πράσινη οικονομία τι σημαίνει. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα και στο Ρίο είναι αυτό πρόβλημα. Γιατί μερικές φορές φαίνεται οι στόχοι που προτείνουμε είναι οι στόχοι που προτείνονται από όλα μέρη του κόσμου, στον τρίτο κόσμο και πάντα κολλάμε στην υλοποίηση. Πάντως, όταν μιλάμε για αυτούς τους στόχους που εμείς προτείνουμε, τους στόχους αυτούς τους έχουμε θέσει πρώτα στους εαυτούς μας. Και οι υποανάπτυξη χώρες βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Άρα πρέπει να τροποποιήσουμε τις δικές μας οικονομικές πολιτικές και να γίνει κατανοητό ότι η πράσινη οικονομία είναι μια κάπως διαφορετική ιστορία από αυτή την οποία είχαμε κατά το παρελθόν. Έχει να κάνει με την δικιά μας την αλλαγή, ακόμα και αν δεν κυριαρχούμε στις διαδικασίες. Συγχρόνως βέβαια, η πράσινη οικονομία είναι και μια έννοια που λέει ότι σταματάει, γίνονται ριζικές αλλαγές και ότι όλα θα πρέπει να σταματήσουν. Άρα, όχι, δεν είναι έτσι. Η οικονομία που δεν ήταν πράσινη μέχρι τώρα έχει δείξει και τα όρια της όσον αφορά την ανάπτυξη. Και γι' αυτό αρχίσαμε να μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη, γιατί λαμβάνει υπόψη της και άλλα πράγματα και το κοινωνικό επίπεδο και το περιβάλλον αλλά και την ε, οικονομική ευρωστία. Πράγματα τα οποία πρέπει να αποτελέσουν μέρος μιας μελλοντικής οικονομίας η οποία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε με ευημερία και που θα ανταποκρίνεται στις σημαντικές προκλήσεις που έχουμε σήμερα μπροστά μας και που βάζουν όρια στην ανάπτυξή μας, στην ανάπτυξη δηλαδή αυτής της μη πράσινης οικονομίας που είχαμε κατά το παρελθόν. Όσον αφορά τώρα την αποψήλωση των ε, δασών, και αυτό είναι κάτι το οποίο συζητάμε με την Βραζιλία και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε ικανοποιητικές λύσεις σύντομα. Είναι ένα εσωτερικό θέμα που παρακολουθούμε πάντως στενά. Για τα ύδατα νομίζω ότι μίλησα για την ισορροπία που πρέπει να υπάρχει. Απάντησα στην κυρία Μαζοκούκοβιτς. Έχετε δίκιο βέβαια ότι πρέπει να τα λάβουμε αυτά υπόψη μας. Το μόνο που θα είχα να προσθέσω σε αυτό που είπατε εσείς είναι ότι για πολλά από τα θέματα που συζητάμε όσον αφορά αυτή την αποδοτικότητα των πόρων είναι ότι όλα αυτά ε, μας δείχνουν ακριβώς την εικόνα του πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη σχετική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στο μέλλον υπάρχει τεράστια εξάρτηση. Οι πρώτε ύλε, ε, οι τιμέ του ανεβαίνουν στα ύψη. Δεν πρέπει να το αγνοούμε αυτό. Γιατί αν το αγνοούμε, τότε μπαίνουμε σε μια κατεύθυνση από την οποία θα υποφέρει πάρα πολύ η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Για νέα προϊόντα, τα οποία θα χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια, λιγότερο νερό, που θα ανακυκλώνονται κτλ. Όλα αυτά οικονομικά έχουν νόημα. Και γι' αυτό και σας διάβασα τη διατύπωση αυτή πριν του πώς ε, βλέπουν οι επιχειρήσεις στο μέλλον τους. Η ισορροπία αυτή υπάρχει λοιπόν. Εδώ έχω τρεις σελίδες ακόμα. Πρόεδρος, έχω πέντε συναδέλφους που έχουν ε, ζητήσει ακόμα το λόγο που τον έχω ζητήσει από την προηγούμενη εβδομάδα και άλλοι δύο ζήτησαν σήμερα το λόγο. Αυτοί οι επτά λοιπόν μπορούν από ένα λεπτό καθένα, μία ερώτηση ο καθένα και να απαντήσετε μετά. Ε, όλα είναι δυνατά, λέει ο Επίτροπο. Ωραία. Κύριε Επίτροπο, έχετε το λόγο. Ωραία και θα πούμε και μερικά πράγματα για την εφαρμογή. Communication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 την 7η Μαρτίου είχαμε μια ανακοίνωση ε, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τα αναχρονισμένα εργαλεία. Ε, επίσης πρέπει να πω ότι εκμονήσαμε μελέτες οι οποίες ε, δείχνουν ότι, στον καλό, ότι η καλή εφαρμογή έχει οδηγήσει σε μεγάλες αποταμιεύσεις. Η σωστή εφαρμογή και η σωστή υλοποίηση των οδηγιών θα μπορούσαν να οδηγήσουν οδηγήσουν σε δημιουργία 400.000 θέσεων εργασίας και επίσης θα οδηγήσουν σε ένα σημαντικό οικονομικό ε, όφελος. Ε, θα πρέπει εδώ να υπενθυμίσουμε ότι το κόστος της μη εφαρμογής είναι πάρα πολύ μεγάλο και βεβαίως εδώ δεν ε, υπολογίζω και την επίπτωση στην υγεία. Στην ανακοίνωση αναφερόμαστε σε δύο στοιχεία όσον αφορά το πρώτο, δηλαδή την γνώση. Οπωσδήποτε θα πρέπει να διαρθρώνεται και να παρουσιάζεται καλύτερα η πληροφόρηση έτσι ώστε να είναι καλύτερη η εφαρμογή της. Βεβαίω, ε, θα πρέπει ταυτόχρονα να προωθήσουμε το e-government, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Κατά αυτήν την έννοια εμείς ε, ε, λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρης χρήση των εργαλείων τα οποία μοιραζόμαστε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με ad hoc συλλογή πληροφοριών. Επίσης, να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά ζητήματα εφαρμογής μεταξύ των κρατών μελών. Και επίσης, να είμαστε οι ίδιοι πιο διαφανείς και να βελτιώσουμε ε, και την ε, ε, δυνατότητα αναφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει ταυτόχρονα καλή αξιολόγηση των πληροφοριών. Θα πρέπει να έχουμε σωστές πληροφορίες όσον αφορά την επιβολή των ε, Τη νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Δεύτερον, όσον αφορά τώρα την ε, ανταπόκριση που είναι το δεύτερο στοιχείο, θέλουμε να έχουμε ένα καλό σύστημα εποπτείας το οποίο θα βασίζεται στις παρούσες ε, συστάσεις όσον αφορά την, τις υφιστάμενες δομές αλλά και τις μελλοντικές δομές εποπτείας. Ε, ενδεχομένως ε, θα πρέπει να ε, δοθούν νέες αρμοδιότητες Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή θα γίνονται περισσότερες επιθεωρήσεις από τα κράτη-μέλη ή κοινέ επιθεωρήσεις. Θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και ε, τα παράπονα των, και οι προσφυγές ε, των πολιτών ε, και όσες προσφυγές φτάνουν στα δικαστήρια καθώς επίσης να βοηθούνται οι αρμόδιες αρχές με μια αποτελεσματικότερη και γενικότερη έποψη όλων των προσφυγών καθώς επίσης και σωστή χρήση του μηχανισμού αντιμετώπισης και φιλικού κύδια διακανονισμού ε, των ε, προσφυγών. Ε, κατά αυτή την έννοια εμείς λέμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη δικτύωση μεταξύ του δικαστικού προσωπικού, των δικηγόρων και όσων ασχολών των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα καλύτερο κατόφλιο εμπιστοσύνη. Επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει οι δικές αρχές οι οποίες θα αφορούν τα συγκεκριμένα προβλήματα των κρατών μελών να δημιουργηθούν. Αυτό ίσως είναι πιο ε, πιο ε, ε, καινοτόμο και πιο επαναστατικό γιατί λέμε στην ουσία εδώ όταν έχετε συγκεκριμένα προβλήματα τότε εσείς από μόνοι σας μπορείτε να προτείνετε την δυνατή λύση και μετά εμείς να βοηθήσουμε έτσι ώστε να ξεφύγουμε από αυτό το αδιέξοδο. Πολύ ωραία. Μία ερώτηση, λοιπόν μάλλον ο κάθε ομιλητής μία ερώτηση και δεν θα ξεπερνάει το ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση πολύ σύντομη, αλλά που για μας που εκλεγόμαστε στην Νότια Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι κοκοφίνικες έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Ε, έχουμε πρόβλημα με τον κόκκινο ξύριχο που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στους ε, φοινικές μας. Έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ειδικό νομοθετικό εργαλείο ε, έτσι ώστε να καταπολεμηθούν τα ιδιαίτερα παρεμβατικά είδη και αυτό σε τον ορίζοντα του 2020. Ποια θα είναι, ποιος θα είναι ο συντονισμός ανάμεσα σε αυτό το νέο εργαλείο και το σύστημα της φυτογενομικής προστασίας στο το οποίο αναθεωρεί αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια θα είναι η διάρθρωση των δύο κατά αυτή την έννοια. Ε, κυρία Δεν πρόκειται για νέο ζήτημα. Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να έχουμε και καλύτερους ορισμούς και καλύτερη έρευνα, περισσότερη έρευνα κτλ. Ε, επίσης υπάρχει και μία αρχή που λέει ότι ε, μπορούμε να παίρνουμε μέτρα έστω και αν δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι. Ε, και τι θα κάνετε όσον αφορά ε, θέματα παρεμβατικών ειδών και ζώων στην επόμενη θητεία. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για το θέμα της εφαρμογής. Νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν πρόβλημα εφαρμογής, γιατί οι διαδικασίες που χρησιμοποιούμε στην Ένωση για να εφαρμόζουμε τα νομοθετήματά μας σημαίνουν μάλλον και για να εγκρίνουμε τα νομοθετήματά μας σημαίνουν ότι υπάρχουν πολλοί συμβασμοί κάτι το οποίο δεν ικανοποιεί τους ανθρώπους γι' αυτό κολλησιεργούν θα πρότεινα λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά αντί να φτιάχνουμε διάφορες ε, υπηρεσίες αστυνόμευσης και επιβολής να δούμε πώς καταλήγουμε στα νομοθετήματα, να δούμε πώς θα μπορούσαν να απλοποιηθούν και να γίνονται ευρύτερα αποδεκτά, για παράδειγμα. Το Φεβρουάριο 2010 δημοσίευσε μια ανακοίνωση για την αρχή της πρόληψης, όπου είπατε ότι θα πρέπει οποιοδήποτε νομοθέτημα να, ε, ε, ε, οποιοδήποτε νομοθετήματος να προηγείται μελέτη επιπτώσεων. Εφαρμόζετε εσείς ε, αυτές τις διατάξεις, αυτή τη διάταξη για όλα τα νομοθετήματα. Είναι ανεφάρμοστα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κορτίνεθ. Ευχαριστώ. Δύο-τρία άλλα θεματάκια θέλω να θίξω εγώ. Ένα από αυτά είναι το εξή. Για το θέμα των υδάτων. Έχω την εντύπωση ότι όλη την περιβαλλοντική πολιτική την βασίζουμε στις προσφυγές. Ε, μην ξεχνάμε τι γίνεται με το Natura 2000. Πάντα υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις εκεί χωρίς να μπορεί να εφαρμοστεί κάθε απόφαση. Ρωτάω λοιπόν, δεν θα έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και να ξέρουμε ποιες ακριβώς είναι αποφάσεις με τα ψηφιακά, με το European Space, με τα συστήματα που έχουμε καθημερινά. Δεν θα έπρεπε να πετούμε περισσότερη διαφάνεια και να ξέρουμε τι τηρείται και τι δεν τηρείται και από ποιον. Να υπάρχει έλεγχος, όπως και για τα ποτάμια. Δεύτερον, πιστεύω και παραλαμβάνω ότι απομακρυνόμαστε από το θέμα της βιωσιμότητας στο οποίο αναφέρθηκαν διάφοροι και το θέμα των αστικών χώρων. Γιατί η βιωσιμότητα, η εφορία πρέπει να βασίζεται από το χώρο όπου εφαρμόζονται διάφορες διατάξεις, ήδο, κλιματικές αλλαγές. Εγώ δεν βλέπω καμιά αστική πολιτική που να τα λαμβάνει αυτά υπόψη. Τι κάνουμε, ε, φυτεύουμε μερικά δέντρα, μειώνουμε 2-3 βαθμούς την θερμοκρασία και τελείωσε και τίποτα άλλο. Έληξε ο χρόνος σας. Καλή Φαμπρέντ και μετά πώς θα Καλή Φαμπρέντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, όπως γνωρίζετε δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ενέργεια και η απόδοση σε ενέργεια, μας ενδιαφέρει και ο, ο χάρτης πορείας είναι πολύ βασικό και το κοινοβούλιο μας τον έχει υπογραμμίσει πάρα πολύ το θέμα του αερίου σχιστόλιθου. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να κάνει εκθέσεις αντικτύπου για το περιβάλλον στις κατοικημένες περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν έχει προχωρήσει αρκετά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να ικανοποιείται με μία μόνο έκθεση αντικτύπου για ένα μόνο θέμα. Για μας αυτό είναι ένα πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να μας απαντήσει περισσότερο και να μας πει πώς θα φροντίσει να υπάρξει ηγετικός ρόλος σε αυτά. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Πρώτον, για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, η οποία μειώνεται ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντο λέει κατά 2,5% έχει μειωθεί από το 2009. Ενώ οι χώρε μέλη δεν εφαρμόζουν καν τι ίδιε προδιαγραφέ. Τι θα κάνετε λοιπόν για να βελτιώσετε τα πράγματα. Δεύτερη ερώτηση. Ποιότητα του αέρα. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά τα πειράματα που γίνονται για την αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ. Ρώση. Ένα λεπτό, ε. Το κομισάριο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ γιατί προηγουμένως δεν απαντήσατε στις ερωτήσει σας. Γι' αυτό λοιπόν κάνω και μία τρίτη. Μιλάτε για ε, επικαιροποίηση και πληροφόρηση μάλλον των ε, πολιτών. Οι πληροφορίες όμως ε, για την ε, βιομηχανία που ε, χρησιμοποιούν ας πούμε διάφορα αέρια και τα, και τα παράγωγά τους, κυρίως η στρατιωτική βιομηχανία που έχει ιδιαίτερες χρησιμοποιεί ουσίες για τις οποίες δεν υπάρχουν ούτε καν συγκρίσιμα στοιχεία και δοκιμαστικά συγκρίσιμα στοιχεία. Ε, αυτή τη στιγμή λοιπόν τι κάνουμε με τη βιομηχανία η οποία είτε μεταποιεί είτε χρησιμοποιεί αυτά τα ε, στοιχεία. Κύριε Επίτροπε, ξέρω ότι είναι πολύ φιλόδοξο το, προ... το, ενδεχόμενο να απαντήσετε σε όλα, αλλά σας δίνω το λόγο παρόλα αυτά. Ευχαριστώ. Για τα επιθετικά είδη. Ναι. Θα υπάρξει νομοθετική πρόταση φέτος. Ωραία, αυτή ήταν εύκολη, σαφή απάντηση. Είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ε, υγεία και ΣΑΝΚΟ, βεβαίω συνεργαζόμαστε. Είμαστε υποχρεωμένοι. Γιατί είμαστε τμήμα του ίδιου οργάνου και πάντα επιδιώκω συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Οι διαταράκτες ε, των ορμονών. Είπαμε ότι θα αναθεωρήσουμε τη στρατηγική μας αυτή τη στιγμή, αν χρειάζεται. Θα την επανεξετάσουμε και αν χρειαστεί θα την αναθεωρήσουμε. Ήδη παραγγείλαμε μια μεγάλη μελέτη για τα χημικά που διαταράσσουν την ορμονική λειτουργία. Τον Ιανουάριο είδαμε τα αποτελέσματα. Φέτος, νωρίτερα, το μήνα αυτό, υπήρξε μια νέα έκθεση που βασίζεται σε 15 έτη έρευνας και προσπαθεί να δει πώς επηρεάζεται το περιβάλλον, οι άνθρωποι, τα είδη. Θα κάνουμε μια μεγάλη διάσκεψη 11 με 12 Ιουνίου στις Βρυξέλλες για το θέμα αυτό των ε, ενδοκρινικών διαταρακτών. Ελπίζω να συμμετέχουν 200-300 άτομα. Προσπαθούμε να έχουμε μια πλατιά συμμετοχή από διάφορες απόψεις. Σημαντικό βήμα μπροστά αυτό λοιπόν. Και βεβαίως ε, ε, ε, έχουμε και διάφορα νομοθετήματα για το θέμα αυτό που πρέπει να εφαρμόσουμε το 2013. Πρέπει δηλαδή μέχρι τέλος του 2013 η Επιτροπή να προτείνει κριτήρια για να εντοπίζουμε ουσίες που έχουν τέτοιες ιδιότητες διατάραξης στις ορμονικές λειτουργίες και να υπάρξει ένα νέο νομοθέτημα για το θέμα αυτό, ένας νέος κανονισμός. Σωστά τονίσατε ότι οι οδηγίες μας δεν είναι πάντα εύκολο να κατανοηθούν και να εφαρμοστούν. Βέβαια δεν ισχύει πάντα αυτό. Αλλά σίγουρα και εγώ θα συμφωνούσα. Πρέπει στόχος μας όταν ε, εκπονούμε προτάσεις πρέπει να είναι και αυτός. Αλλά όπως ξέρετε οι προτάσεις ε, έχουν ε, νομικό χαρακτήρα. Αλλά οπωσδήποτε ε, δεν είναι εύκολο για τους πολίτες να τις καταλάβουν. Είδα τα κολύμβησης. Α, α, ενέργεια, ενέργεια, η ερώτησή σας. Και σχιστολιθικό αέριο με το τωρινό μας πλαίσιο, κανονιστικό πλαίσιο, τα κράτη-μέλη αποφασίζουν εάν θα επιτρέψουν την ε, έρευνα και την παραγωγή αερίου από σχιστολιθικά πετρώματα, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως την νομοθεσία που έχουμε από κοινού εγκρίνει. Ούτως έχει η κατάσταση από νομική άποψη. Πέρυσι η Επιτροπή έκανε μια μελέτη του κανονιστικού πλαισίου για αυτό το αέριο και θεωρεί ότι μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το πλαίσιο για την έρευνα και την παραγωγή σχιστολιθικού αερίου. Συμφωνούμε με το Κοινοβούλιο γι' αυτό. Επίση, αρχίσαμε την εργασία για να αποτιμήσουμε μέχρι το τέλο του 2013, εάν και κατά πόσο, το πλαίσιο αποτίμηση των κινδύνων από την παραγωγή σχιστολιθικού αερίου είναι επαρκέ ή αν θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα ειλικρινά το θέμα αυτό πρέπει να το καταλάβουμε κάπως καλύτερα. Σε αυτή τη φάση εργαζόμαστε έντονα για να συλλέξουμε περισσότερες ε, πληροφορίες, αλλά είναι σαφές ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, που έχουν περισσότερη πείρα από τη χρήση και παραγωγή σχιστολιθικού αερίου προκύπτουν όλο και περισσότερα στοιχεία που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι το περιβαλλοντικό θέμα θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Τέλος. Είδα τα κολύμψη. Οι παραλίες. Έχουν ε, μικρές αλλαγές. Έχουν γίνει μικρές αλλαγές στην ποιότητα από χρόνο σε χρόνο του νερού στις παραλίες. Αλλά αν δούμε τι απόσταση έχουμε διανύσει από τότε που εισήχθη η νομοθεσία για τα θέματα αυτά, Πρέπει να είμαστε περήφανοι. Ε, έχουν σημειωθεί μεγάλες πρόοδοι σε σχέση με το παρελθόν. Βεβαίω, οι διακυμάνσει ε, σημαίνει πως πρέπει να είμαστε πάντα σε επαγρύπνηση. Και αυτό κάνουμε. Και αυτό θα κάνουμε. Για την αποθήκευση του διοξίδιου του άνθρακα. Δεν κατάλαβα. Συνδέεται με θέματα που θα τα λάβουμε υπόψη στις επενδύσεις μας. Αν είναι σημαντικό τμήμα, εγώ πάντα το θεωρούσα, σημαντικό τμήμα την αποθήκευση του διοξίδιου του άνθρακα. Οπωσδήποτε πρέπει να το αντιμετωπίσουμε γιατί πολλέ χώρε σε διάφορα σημεία του κόσμου δεν μπορούμε να αναμένουμε ότι σύντομα και αποτελεσματικά θα περάσουν σε μορφές παραγωγής ενέργεια πιο φιλοπεριβαλλοντολογικές. Γι' αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε είτε μας αρέσει είτε όχι, θα είναι τμήμα της φροντίδας μας. Το θυμάμαι και από την προηγούμενη ενασχόλησή μου, την προηγούμενη ιδιότητά μου. Για τα αέρια με νευροτοξίνες. Δεν ξέρω κύριε Ρώση τίποτα για το θέμα αυτό. Θα απευθυνθώ στις υπηρεσίες μου. Τέλος. Ένα τελικό σχόλιο. Καταλαβαίνω πολλές φορές ε, την ανυπομονησία σας, την απόγνωσή σας για τις βραδίτητες της εφαρμογής. Πιστεύω πως αν ήσασταν θέση μου θα ήσασταν ακόμη πιο ενοχλημένος. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον διάλογο, αυτή την ε, δυνατότητα που μας δώσατε Επίσης ε, για την ε, διάθεσή σας να μείνετε παραπάνω μαζί μας. Είστε πάντα καλοδεχούμενος στην Επιτροπή μας κύριε Επίτροπε. Είμαστε στο ίδιο χαράκομα. Αλλά παρακαλώ η προθεσμία για την υποβολή νομοθετημάτων είναι Μάρτιος του 2013 για το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το διάλογο και την παρουσία σας εδώ. Λοιπόν, μετά αυτόν τον διαρθρωμένο διάλογο συνεχίζουμε. Ηχοστάθμη μηχανοκινήτων οχημάτων. Το επόμενο θέμα μας, εισηγητής, ο συνάδελφος Μύροσλαβ Ούσκι. Και του δίνω το λόγο για να με εισαγάγει το θέμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας περιμένουμε όσοι θέλουν να εγκαταλείψουν την αίθουσα να βγουν και να μείνουν αυτοί που θέλουν να παρακολουθήσουν. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι παρουσιάζει μία λύση προκειμένου να περιοριστεί η χορύπανση στο περιβάλλον μας. Πιστεύω όμως ότι θα ήταν καλό να διευρύνουμε ακόμα περισσότερο και να τροποποιήσουμε λίγο το, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να δώσουμε κίνητρα στην παραγωγή και να πετύχουμε νέα οχήματα με χαμηλά επίπεδα θορύβου. Το επίπεδο θορύβου των οχημάτων οφείλεται βέβαια σε διαφορετικούς λόγους. Είναι ο κινητήρας πρώτα απ' όλα, είναι τα λάστιχα, είναι ο τρόπος οδήγησης, είναι το δόστρωμα κλπ. κλπ. Το πρόβλημα συχνά ε, λύνεται με μια καλή διαχείριση της μεταφοράς που έχει σαν αποτέλεσμα τα φορτηγά, τα μεγάλα, τα βαρέα οχήματα να φεύγουν από τους κύριους άξονες. Θέλω εδώ να αναφερθώ πάντως στην επιφάνεια των δρόμων, στο δόστρωμα που είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί λοιπόν το το... η πρόταση αυτή της Επιτροπής προσθέτοντας ένα σύστημα ταξινόμησης των οδικών αρτηριών έτσι ώστε οι χώρες μέλη να μπορούν πιο εύκολα να ελέγχουν την κατάσταση εκεί, να αξιολογούν το οδόστρωμά τους και έτσι να βελτιώνουν τις επιπτώσεις που έχει αυτό στον θόρυβο των οχημάτων. Υπάρχουν βέβαια διάφορες τεχνικές προδιογραφές που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που μετράμε ε, τον θόρυβο των κινητήρων. Δεν χρειάζεται να μπω στις λεπτομέρειες. Πάντως ε, ο στόχος μας είναι μέθοδοι μέτρησης ικανοποιητικές και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται οι μετρήσεις αυτές που πρέπει να ακολουθεί τις σωστές παραμέτρους. Υπάρχουν οριακές τιμές, υπάρχουν και τέσσερα στάδια εφόσον χρειάζεται να μπορούμε να καταλήξουμε έτσι στην καλύτερη δυνατόν μέτρηση μετά από το τέλος του σταδίου 3. Οι οριακές τιμές έτσι όπως αναφέρονται στο παράρτημα 3 της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελούν ένα βασικό στοιχείο του κανονισμού. Είναι θέμα συνομοθετών. Συνεπώς, συμφωνώ με την πρόταση που λέει ότι η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει ε, τέτοιες ε, τεχνικές προδιαγραφές μέσω ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων. Τα υπόλοιπα πρέπει να γίνονται με συναπόφαση σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή σας και στην τροπολογία 19. Τελικά αποφάσισα να αποσύρω την τροπολογία αυτή γιατί αναγνωρίζω η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι προτιμότερη. Όσον αφορά τώρα την υποχρεωτική σήμανση ε, για το ευρύ κοινό. Εδώ δεν είναι ξεκάθαρο το τι ενδιαφέρει τελικά τον καταναλωτή, αν είναι πιο πολύ ο θόρυβος έξω από το αυτοκίνητο ή μέσα στο όχημα. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να έχουμε μια μελέτη αντικτύπου επ' αυτού, γιατί είναι διαφορετικά τα πράγματα στη μία και στην άλλη περίπτωση. Περιμένω τις δικές σας παρατηρήσεις και σχόλια. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Um, that Ευχαριστώ κύριε σκιώδες εισηγητές τώρα. Πρώτος από πλευράς έλκο κύριο Στατάρελα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μύροσλαβ για την εργασία του αλλά και για την συνεργασία που είχαμε στα πλαίσια της εκπόνησης αυτού του εγγράφου ε, και της προηγούμενης συζήτησης. Θα ήθελα να πω ε, την άποψή μου και ε, να παρουσιάσω εντάχει κάποιες τροπολογίες. Όπως είπα και σε κάποιους άλλους σκιώδεις, συναδέλφους θεωρώ ότι αυτό το ζήτημα δεν θα πρέπει να έχει μονάχα ε, ε, κάθετη αλλά και ε, καλύτερα ακόμα οριζόντια προσέγγιση. Δεν μπορούμε δηλαδή να μιλάμε μονάχα για αυτοκίνητα και για θόρυβο αν δεν αναφερθούμε και στις υποδομές και στα ελαστικά. Όσον αφορά τα ελαστικά ε, υπάρχει νομοθεσία, αλλά όσον αφορά ε, τους δρόμους και τις υποδομές, ε, πολλά μπορούν να γίνουν ακόμα και θα προς αυτό κάνω έκκληση για το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις οι οποίες όσον αφορά την ταξινόμηση των οχημάτων τα εξέφρασε ήδη ο συνάδελφος με πολύ ικανοποιητικό τρόπο, επομένως με βρίσκει σύμφωνο. Πρόθεσή μου είναι να στηρίξω την ιδέα της δημιουργίας μιας νέας κατηγορίας ε, που θα ε, αφορά ε, τα αυτοκίνητα μικρού όγκου, small volume car που αποτελούν το 0,03% της παραγωγής και που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ειδική κατηγορία με ειδική νομοθεσία. Επίσης, συμφωνώ απολύτως με τις τροπολογίες που υπέβαλε ο εισηγητής όσον αφορά τα, ε, τις δοκιμές μέτρησης, αλλά όσον αφορά αυτή, αυτές τις επισημάνσεις στις οποίες αναφέρεται είμαι λίγο διστακτικός. Είναι προφανές ότι αυτές οι ενδείξεις

μπορούν να χρησιμεύσουν στον ε, καταναλωτή. Αλλά όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως υπάρχει μία σύγχυση σχετικά με τον θόρυβο. Αν θα είναι ο θόρυβος έτσι όπως ε, τον ε, καταλαβαίνουν ο οδηγός και οι υπόλοιποι επιβάτης ή ο θόρυβος έτσι όπως τον ακούν και τον αντιλαμβάνονται όσοι είναι έξω από το αυτοκίνητο. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να επιληθεί αφορά τώρα την εναρμόνιση των συστημάτων αξιολόγησης αυτού του θορύβου ε, και αυτό το σύστημα θα πρέπει να συζητηθεί γιατί μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες ε, παρανοήσεις και ενδεχομένως και παρεξηγήσεις. Πιστεύω ότι το ζήτημα αυτό μπορούμε να το διαχειριστούμε καλύτερα, ε, ίσως στην Επιτροπή ΙΜΚΟ, με ένα ειδικό, ε, ε, με ένα ειδικό φάκελο που θα ασχοληθεί ακριβώς με αυτές τις λεπτομέρειες και δεν χρειάζεται εμείς να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες και βεβαίως ε, χρειάζεται και επίπτωση, αξιολόγηση συγγνώμη, επιπτώσεων. Επίσης, όσον αφορά την κατηγοριοποίηση η οποία οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει λίγο πιο εύκολη, κυρίως για τα ε, μικρά οχήματα, λιγότερο των 50 κιλοβατόρων. Επίσης, να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα άλλο ζήτημα, δηλαδή το θέμα των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος που μας απασχολεί ήδη και σε άλλες περιπτώσεις. Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η αποθήκευση έστω και ενός τμήματος του ε, κινητήρα ε, μπορεί να σημαίνει ε, μεγαλύτερη, μεγαλύτερες εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακος. Ο εγκυβωτισμός, συγγνώμη. Ε, λοιπόν, θεωρούμε ότι η έκθεση αυτή είναι εξειδικευμένη, αναφέρεται πολύ σωστά στα ζητήματα ε, τα οποία ε, περιλαμβάνει ε, και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα επί του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Ταταρέλα. την Μέρκης εξ ονόματος των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ. Θα αρχίσω με ευχαριστίες για την καλή συνεργασία που είχαμε με τον εισηγητή που κατάφερε να συμβιβάσει τις διάφορες απόψεις. Πράγματι είναι για μια τεχνική υπόθεση αυτή. Μιλήσαμε και με τον Επίτροπο Ποτότσκι και το θέμα του επίπεδου θορύβου είναι ένα στοιχείο που επηρεάζει πάρα πολύ την καθημερινή μας ζωή, αλλά προκαλεί μάλιστα και πολλές ε, ασθένειες ή τέλος πάντων είναι υπεύθυνο για διάφορες ασθένειες σε ένα βαθμό, αν μη τι άλλο. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε ένα αποδεκτό επίπεδο θορύβου από την κυκλοφορία και από τα οχήματα. Είναι κάτι πολύ βασικό για την ευημερία μας και για την αποφυγή διαφόρων ασθενειών. Πιστεύω επίσης είναι και η άποψη του κυρίου Ούσκη, με την οποία συμφωνώ και εγώ, ότι είναι θέμα κατασκευής του οχήματος. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που επηρεάζουν το θόρυβο, όπως είπαμε και εμείς, και το δόστρωμα και τα λάστιχα και οδήγηση και όλα. Οπότε το ερώτημα είναι, πού βρισκόμαστε σήμερα, τι ακριβώς κάνουμε, κοιτάμε όλα αυτά τα θέματα ή μήπως τελικά ε, κοιτάζουμε μια οδηγία που έχει να κάνει ε, με τον θόρυβο των οχημάτων, δηλαδή τον θόρυβο που κάνει ο κινητήρας του οχήματος και τίποτα από όλα τα υπόλοιπα που επηρεάζουν τελικά τον θόρυβο από τα οχήματα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε όλα και όχι μόνο τον θόρυβο που βγαίνει από το όχημα να δώσουμε συνέχεια και στα άλλα ε, θέματα, δηλαδή εν ώψη της οδηγίας για την χορύπανση. Και έχω και μερικά άλλα πράγματα που θέλω να αναφέρω. Πιστεύω ότι η πρόταση του εισηγητή έχει αποδυναμωθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοίμασε μια καλή πρόταση. Το 65% των οχημάτων, από ό,τι φαίνεται, ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε εγώ δεν βλέπω γιατί πρέπει να αποδυναμώσουμε τις τιμές αυτές περισσότερο. Τη συζήτηση την κάναμε αντίστοιχα και για τις προδιαγραφές του οξυδίου του άνθρακα. Μην ξεχνάμε ότι, όπως είπα, πολλά οχήματα ανταποκρίνονται ήδη τι χρονό και τι περιθώριο πρέπει να δώσουμε στο υπόλοιπο 35%. Ένα άλλο θέμα που μου απασχολεί είναι οι δοκιμές που γίνονται. Η χαμηλότερη τιμή είναι αυτή η οποία τελικά θα ισχύσει. Αυτή είναι η πρόταση. Γιατί εγώ νομίζω, αν δω την σχετική τροπολογία, η οποία βασίζεται σε παλιότερα αποτελέσματα δοκιμών και όχι στις νέες ε, δοκιμές, έχω πολλές αμφιβολίες. Κατά τα άλλα, ευχαριστώ τον εισηγητή που μίλησε και για την ακρόαση για την ηχοστάθμη. Και αυτό που με ενδιαφέρει επίση είναι και η σήμανση. Δηλαδή ότι ο καταναλωτή να μην ξέρει μόνο τι γίνεται με το διοξίδιο του άνθρακα, με την ενέργεια κτλ. για το όχημα που θα αγοράσει, αλλά να είναι ενήμερο και για τα επίπεδα θορύβου που προκαλεί το όχημα το οποίο πρόκειται να αγοράσει. Ευχαριστώ πολύ και για τι θέσει μου, τι οποίε δέχτηκε ο συγητή επόμενος ε, συνάδελφο, ο κύριο Κράμερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την ε, καλή εργασία που επετέλεσε. Νομίζω ότι διόρθωσε ορισμένα σημεία που στην πρόταση της Κομισιόν προκαλούσαν μεγάλα ερωτηματικά για την ε, ταξινόμηση για παράδειγμα. Πρότεινε πράγματα που δεν ισχύουν πλέον εδώ και καιρό. Γιατί λοιπόν η Κομισιόν προσπαθεί να ρυθμίσει τα οχημάτων που δεν υφίστανται πλέον, δεν πουλούνται. Θέλω να υπενθυμίσω ότι οι νόμη μας πρέπει να είναι σε αρμονία με τον κύκλο παραγωγής. Ορισμένα οχήματα δεν είναι δυνατόν να ζητάμε να δημιουργηθούν επειδή έχουμε νόμους εμείς που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Πρέπει να καταλαβαίνουμε πώς και να συνεργαζόμαστε με την παραγωγή. Βεβαίως. Πρέπει να μειωθεί ο ήχος από τα, ο θόρυβος από τα οχήματα, γιατί η επιβάρυνση από τον θόρυβο των οχημάτων, κυρίως ε, στις πόλεις, είναι μεγάλος. Έχω μία ερώτηση για το τέταρτο σημείο. Δεν ξέρω τι έννοια έχει να έχουμε μακροπρόθεσμους στόχους σε ένα νομοθέτημα για 14 ή 16 χρόνια. Πιστεύω ότι πριν αναφέρει κανείς ε, αριθμούς θα πρέπει να κάνει την ε, επανεξέταση και την μελέτη των επιπτώσεων. Από ό,τι διάβασα εγώ τουλάχιστον, οι στόχοι αυτοί, οι τόσο μακροπρόθεσμοι, δεν είναι καθόλου εφικτοί ε, αν δεν αλλάξουμε και άλλους νόμους, για παράδειγμα για τα ελαστικά. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η σωστή μέθοδος. Ε, τόσο μακροπρόθεσμη εφαρμογή θα έπρεπε να καταργηθεί. Το είπαν ε, και όλοι οι συνάδελφοι. Το θόρυβο δεν τον προκαλούν μόνο τα οχήματα, τον προκαλούν και τα ελαστικά, τα οδοστρώματα, άρα είναι θέμα συνολικά της πολιτικής συγκοινωνιών και μεταφορών. Πρέπει να κάνουμε έναν ε, νόμο που να αφορά την, ε, σε αυτή τη φάση την ε, έγκριση διαφόρων τύπων οχημάτων. Τώρα, για παράδειγμα, η κατάταξη των οδοστρωμάτων, να τη συζητήσουμε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή εδώ. ετικέτες για το θόρυβο τώρα δεν ξέρω τι περισσότερη, τι προστιθέμενη αξία δίνει στο καταναλωτή. Έχω την εντύπωση ότι σε διάφορα σημεία μέσω ενωσιακών νομοθετημάτων κάνουμε κάτι υπερβολικό. Ε, ξέρω ότι θα υπάρξει οδηγία για την ετικετοποίηση των ελαστικών. Γιατί πολλοί δεν είναι σίγουροι τι περισσότερα στοιχεία, τι έννοια έχει η παροχή όλων αυτών των στοιχείων στον ε, καταναλωτή. Τι θα καταλάβει από όλα αυτά τα στοιχεία. Θα ήμουν σε αυτήν ε, την σήμανση των ελαστικών να την αποδεχθώ. Αν είμαστε κάπως πιο ρεαλιστές όσον αφορά την προσαρμογή στον ε, τρόπο παραγωγής των οχημάτων στο σχέδιο της Κομισιόν μιλάμε για ελάχιστες ε, απαιτήσει για τα ηλεκτρικά οχήματα. Ρώτησα γιατί το αναφέρουμε αυτό εδώ. Εδώ μιλάμε για μια οδηγία για τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και για τη μείωση των ανεπιθυμήτων επιπτώσεων στην υγεία. Οι ελάχιστες ε, προδιαγραφές θορύβου των ηλεκτρικών οχημάτων είναι θέμα οδικής ασφάλειας. Είχα πάει πριν από λίγο καιρό στην Στουτγάρδη και είδα διάφορες δοκιμές ε, ηλεκτρικών οχημάτων ε, στο κέντρο της πόλης. Πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, θα μπορούσε να μας απασχολήσει. Αλλά για το θόρυβο των οχημάτων αυτών ένα είναι σημαντικό. Όλους αυτούς τους μήνες που γίνονται αυτές οι δοκιμές δεν υπήρξε ούτε μία περίπτωση ούτε μία περίπτωση όπου να έχουν υψηλό θόρυβο, να παράγουν υψηλό θόρυβο αυτά τα οχήματα. Είναι σχεδόν αθόρυβα. Τώρα ελάχιστες λοιπόν προδιαγραφές για το θόρυβο των ηλεκτρικών οχημάτων. Ας εξετάσουμε αν υπάρχει κίνδυνος. Από ποια στιγμή ένα όχημα μπορεί να είναι υπερβολικά ήσυχο και αυτό να δημιουργεί κίνδυνο. Είναι θέμα οδικής ασφάλειας νομίζω και όχι θέμα θορύβου. Κατά τα άλλα ελπίζω να υπάρξει συμβιβασμός να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε θετικά το θέμα αυτό, να έχουμε αυτή την οδηγία γιατί είναι καιρός να μειώσουμε τον θόρυβο από τα οχήματα. Πολύ καλή η πρόταση, σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ, ίσως με μια-δυο τροπολογίες για να τη βελτιώσουμε κάπως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όλγα Εγώ μια φορά παραλίγο να με χτυπήσει ένα ηλεκτρικό όχημα ακριβώς γιατί δεν το άκουσα. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Και τώρα συνάδελφος Άιχορτ ε, που αντικαθιστά το Χάτο Χάση. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που δεν είναι εδώ η κυρία Χάση. Θα την εκπροσωπήσω. Κάτι που κάπως μας εκπλήσει όταν βλέπουμε την έκθεση Ούσκι. Μοιάζει να έχει λιγότερες φιλοδοξίες από ότι η Κομισιόν. Εμείς δεν θα θέλαμε να συμβεί κάτι τέτοιο σε αυτή την έκθεση. Άρα πιστεύω ότι η συζήτηση θα είναι ενδιαφέρουσα. Διορθώστε με αν κάνω λάθος κύριε Ούσκη. Πρώτον λοιπόν, ως κοινοβούλιο πρέπει να είμαστε συνεπείς. Όταν κάνουμε μια έκθεση για το 7ο περιβαλλοντικό πρόγραμμα δράσης και λέμε σαφέστατα ότι πρέπει να υπάρχουν μέτρα για να αντιμετωπιστούν, να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για την υγεία από το θόρυβο και μετά περνάμε σε μια τέτοια οδηγία για τα οχήματα και βλέπουμε υποχώρηση. Ενώ μιλάμε πάντα στα περιβαλλοντικά προγράμματα δράσης για φιλόδοξους στόχους, όταν περνάμε στα συγκεκριμένα νομοθετήματα είμαστε επίση αν έχουμε μειωμένε ε, φιλοδοξίες. Από τον Νοέμβριο του 2012 εξάλλου θα υπάρξουν οι ισχυρότερε προδιαγραφέ για την απόδοση των ελαστικών. Να μας πει λοιπόν η Επιτροπή, διότι από ό,τι ξέρω εγώ αυτές οι αυστηρότερε προδιαγραφέ για τα ελαστικά που θα αρχίσουν να ισχύουν τον Νοέμβριο του 2012 τότε θεωρώ ότι θα έχουν επιτευχθεί οι περισσότερες προδιαγραφές της πρώτης φάσης. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε για την πρώτη φάση πολύ πιο φιλόδοξοι από την Κομισιόν. Να την εφαρμόσουμε λοιπόν από το 13 και όχι το 14. Οπότε περνάω στην τροπολογία 21 του εισηγητή που είναι ακόμη λιγότερο φιλόδοξη αναβάλει ακόμη περισσότερο την εφαρμογή της φάσης 1 και 2. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να είμαστε υπέρ ταχύτερων προθεσμιών για τη φάση 1 και φάση 2, δηλαδή 13 και 15 αντί για αυτά που προτείνει η Επιτροπή. Το αυτό ισχύει, και εδώ δεν συμφωνώ με τον κύριο Κράνμερ, γιατί πιστεύω ότι και για πιο μακροπρόθεσμη επένδυση για την ασφάλεια των παραγωγών χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμες προδιαγραφές. Να εισαγάγουμε λοιπόν μια τρίτη φάση με προδιαγραφές για το 2020, ούτω ώστε οι αυτοκινητοβιομηχανίες να ξέρουν τι θα βρουν μπροστά τους ε, μακροπρόθεσμα. Ζωτικό αυτό. Λείπει πιστεύω από την πρόταση του κ. Ούσκη. Ε, δεν λείπει εννοώ ότι δεν είναι τόσο φιλόδοξο και μια ερώτηση στον κύριο Ούσκι για την τροπολογία 22 γιατί προσθέτει το σημείο που λέει ότι θα πρέπει να μειωθεί ο θόρυβος κατά ένα δεσιμπέλ. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Μήπως μπορεί να μας εξηγήσετε. Δεν την καταλαβαίνω. Καταλήγοντας, συμφωνώ με τον κύριο Κράνμερ όταν τονίζει αυτά που τονίζει για τα ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό αποδεικνύει ότι ορισμένες φορές ε, οι πράσινοι συμφωνούν με τον κύριο Κράνμερ. Καλό να το διαπιστώνουμε και αυτό που και που. Αυτοί ήταν οι σκιώδεις ηγητές. Άνια άμα... Α, έφυγε. τούτα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μία διάσταση που απουσιάζει από τη συζήτηση είναι το γεγονός ότι αν καταφέρουμε να μειώσουμε το θόρυβο των οχημάτων, θα είναι πολύ σημαντικό αυτό και για την ανάπτυξη των πόλεων. Διότι σημαίνει ότι μπορείς σε περισσότερη μία στις πόλεις όπου υπάρχουν υποδομές, ε, να έχουμε δημόσιες μεταφορές, κάτι το οποίο μας κάνει πιο αποτελεσματικούς στην ε, διαχείριση των μεταφορών. Αν όμως δεν μειώσουμε το θόρυβο από τις μεταφορές, τότε όλο και περισσότεροι χώροι κοντά στις πόλεις θα γίνονται ακατοίκητοι και θα πρέπει να πληρώνουμε περισσότερα λεφτά για μεταφορές του κόσμου. Συνεπώς απόσβεση θα γίνει πολλαπλώς γιατί θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ καλύτερα τις πόλεις μας και τις υπηρεσίες των πόλεων. Άρα λοιπόν αυτή την πτυχή πρέπει να την λάβουμε υπόψη μας όταν πάρουμε την απόφαση. Μην μειώνουμε λοιπόν τις φιλοδοξίες μας ε, βάσει στραβών επιχειρημάτων, να νομίζουμε ότι κερδίζουμε χρήματα ενώ τελικά ο λογαριασμός απλώς αλλάζει χέρια, πηγαίνει σε όσους χρησιμοποιούν τις ε, δημόσιες μεταφορές ή επειδή ανακάζει το κόσμος να απομακρύνεται από τις πόλεις και να ζει μακριά για να έχει περισσότερη ησυχία. Να τα έχουμε υπόψη μας όλα αυτά λοιπόν όταν θα αποφασίσουμε. Ευχαριστούμε. Τώρα. Βάση Κέρπα, ευχαριστώ. Με συγχωρείτε επειδή υπήρξε μια αναβολή. Είχα μια άλλη δουλειά. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή κύριο Ούσκι για την ε, καλή πρότασή του. Ως εισηγήτρια στην Ίντα συνεργάστηκα μαζί του και θα ήθελα να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να ανταλλάξουμε απόψεις. Εάν η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει κάποια σημεία που είναι σημαντικά για τους καταναλωτές, για παράδειγμα η σήμανση, στην οποία θα επανέλθω. Χαιρετίζω λοιπόν την πρόταση. Είναι σημαντικό θέμα για την προστασία της υγείας, πάλι για τα αυτοκίνητα, αλλά δεν είναι θέμα εκπομπών, αλλά είναι θέμα βλαπτικών αποτελεσμάτων. Θέλουμε να μειώσουμε το θόρυβο και για λόγους προστασίας της υγείας των οχημάτων. Έχω κάποιες προτάσεις να κάνω από πλευράς προστασίας του καταναλωτή. Το θέμα σήμανση λοιπόν, ο κύριος Ούσκι το ανέφερε και ο κύριος Ταταρέλα, σημαντικό είναι να ενημερώσουμε τους καταναλωτές τι θόρυβο κάνει το αυτοκίνητο γιατί μπορεί να αλλάξει την άποψή του για το τι θα αγοράσει. Αφορά τον πολίτη ως καταναλωτή αλλά αφορά και τα μεσαία στρώματα. Υπάρχουν για παράδειγμα ήδη προγράμματα στην Ολλανδία όπου είναι πολύ σημαντικό τι θόρυβο κάνει το αυτοκίνητο διότι υπάρχουν προδιαγραφές ποια αυτοκίνητα μπορούν να εισέλθουν σε ορισμένες περιοχές των πόλεων. Για παράδειγμα, σε περιοχές ε, όπου κατοικούν οι άνθρωποι, οπότε ορισμένα οχήματα που κάνουν ε, μεταφορές ε, εμπορευμάτων μπορούν να μπουν μόνο από ένα επίπεδο ήχου και κάτω. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Μιλάμε για τον εξωτερικό θόρυβο, για τον εξωτερικό θόρυβο των οχημάτων. Γιατί σε αυτό το νομοθέτημα μας ενδιαφέρει, και ο... μας ενδιαφέρει κυρίως ο εξωτερικός θόρυβος. Γενικά είναι ενδιαφέρον να υπάρχει ενημέρωση του καταναλωτή ως κοινοβούλιο, είναι σημαντικό να την στηρίξουμε, γνωρίζοντας βέβαια ότι δεν είναι μόνο θέμα αυτού του νομοθετήματος, θα καλέσουμε την Κομισιόν να μας κάνει και πρόταση αλλού. Δεν είναι η κατάλληλη ευκαιρία τώρα, αλλά κάνουμε λοιπόν την παράκληση της Κομισιόν να μας πει πώς θα διαρθρώσει συνολικά την νομοθεσία για το θέμα αυτό, αλλά να περιλαμβάνεται ως στοιχείο αυτό είναι σημαντικό για τους καταναλωτές. Και είναι σημαντικό και για μας από πλευρά εσωτερική αγοράς και προστασία των καταναλωτών. Επίσης είναι σημαντικό ότι αναφέρονται διάφορες κατηγορίες. Βεβαίως είναι σημαντικό να υπάρξει νέα διαφοροποίηση. Η πρόταση της Κομισιόν είναι πεπαλαιωμένη. Πρέπει να υπάρξει νέα κατηγοριοποίηση που να ανταποκρίνεται στις νέες κατηγορίες οχημάτων. Για ορισμένες κατηγορίες ε, οχημάτων μπορεί να είναι κανείς πιο φιλόδοξος, για άλλες πιο μετροπαθή σε σχέση με την Κομισιόν. Και εγώ από πλευράς ε, ίντα έχω εργαστεί πολύ, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε μια νέα πρόταση που να είναι όντως όφρον για τον κατάλογο των οριακών τιμών και με χαρά θα συνεχίσω να συνεργάζομαι για τις σημεία πρέπει να είμαστε κάπως πιο πραγματιστές από ό,τι είναι τώρα η πρόταση της Επιτροπής και επίσης να πω στον συνάδελφο Μέρκης που είπε ότι 90% των οχημάτων ήδη πληρούν τις προδιαγραφές της φάσης 1 ναι αλλά αν ε, κάνουμε πιο αυστηρές τις προδιαγραφές τότε θα μειωθεί αυτό το ποσοστό και αυτό το περίπου 40% επίσης κάπως με κάποιο τρόπο να ανταποκρίνονται στις τιμές, διότι αν δεν ανταποκρίνονται τότε συνολικά ο στόλος των οχημάτων δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να συνεχίσει να κυκλοφορεί, γιατί κάποια δεν θα επιτρέπονται. Ε, δεν θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να παραμείνουμε ρεαλιστές. Τελευταίο σημείο. Βεβαίως να υπάρξει σταδιακή εισαγωγή των ε, μέτρων αυτών για τα γιοταχή και για τα φορτηγά, διότι έχουν άλλο κύκλο ζωής. Βεβαίως να βάλουμε μακροπρόθεσμους στόχους, ούτω ώστε και για τους παραγωγούς να υπάρχει προγραμματισμός και ασφάλεια προγραμματισμού. Συμφωνώ με τον Σνάλφο Ούσκι πρέπει να συμπεριληφθεί και ρήτρα αναθεώρηση γιατί πρέπει να μα απασχολήσει περισσότερο για το θέμα αυτό. Αλλά για του συναδέλφους που θέλουν να είναι πιο φιλόδοξοι τότε θα έχουν την ευκαιρία μακροπρόθεσμα μέσω αναθεώρησης να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι. Ίσως αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει βάση συμβασμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βάσκερμπερ. Έχουμε έναν προσκεκλημένο εδώ από την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή, τον κύριο Χανκροάρη και αν δεν έχει κανείς αντίρρηση θα ήθελα να του δώσω το λόγο για δύο λεπτά. Είναι εισηγητή για το θέμα αυτό στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Παρακαλώ, ούτω ώστε από πλευρά Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σύντομα να μα παρουσιάσει την άποψη του θεσμικού οργάνου αυτού. Δεν υπάρχουν αντίρρηση, παρακαλώ. Πρέγκο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Δύο λεπτά έτσι ώστε συνοπτικά να αναφερθώ στη γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής μας. Ε, θα είναι πολύ σύντομη η επεξήγησή μου και θα πω δύο λόγια λοιπόν για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Η Επιτροπή μας, η οποία ενέκρινε τον ε, Απρίλιο, πριν από ένα μήνα δηλαδή, ε, στη, την, τη γνωμοδότηση αυτή στηρίζει την μείωση της ε, της ηχοστάθμης των μηχανοκίνητων ε, οχημάτων, έτσι όπως παρουσιάζεται εδώ. Όμως πρέπει να γνωρίζει κανείς ότι ε, και στην προκείμενη περίπτωση δεν είχαμε ε, ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ε, το άκουσα και αυτό προηγουμένως ε, και είπαμε ότι θα πρέπει ε, να επιτύχουμε τη μείωση της συγχωρήπανσης μέσω της μέτρησης βεβαίως αλλά και μέσω του ελέγχου των ελαστικών, του οδοστρώματος κτλ. Γιατί είναι πολλοί οι λόγοι που γίνονται ε, πιο θορυβόδη οχήματα. Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε ολοκληρωμένη προσέγγιση, γιατί ποτέ ε, δεν θα καταφέρουμε να ε, κατεβούμε κάτω από τον θόρυβο κύλησης των ελαστικών στο δρόμο και αυτό ισχύει και για τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Δεν θα πω περισσότερα σε αυτό το θέμα. Εμείς έχουμε ε, υποβάλει και κάποια άλλα ζητήματα. Μερικά αναφέρθηκαν και εδώ. Το ένα είναι η αναθεώρηση της ε, κατηγοριοποίησης. Ε, γίνεται μια πρόταση τροποποίηση των ιστορικών κατηγοριών έτσι όπως είχαν καθοριστεί το 1985 και εμείς υπογραμμίσαμε το πρόβλημα αυτό αναφορικά και κυρίως ε, με τα αυτοκίνητα One πόρα αυτοκίνητα. Και είπαμε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα είναι εύκολο να αλλάξει η νομοθεσία. Δεύτερον και πιο σημαντικό, ε, το χρονοδιάγραμμα της πρότασης η μείωση θα πρέπει να προέλθει μέσα από πολύ σημαντικές ε, ε, και δύσκολες διαρθρωτικές αλλαγές. Αυτό που προτείνουμε στη δική μας γνωμοδότηση είναι ενδεχομένως να τροποποιήσουμε ε, το χρονοδιάγραμμα ε, και αυτό θα γίνει εάν αφαιρέσουμε την πρώτη φάση που κατά την άποψή μας δεν θα ε, οδηγήσει σε ε, ουσιώδεις βελτιώσεις ή τροποποίησεις. Να εστιάσουμε δηλαδή απευθείας στο τελικό αποτέλεσμα στο οποίο συμπίπτουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μην έχουμε λοιπόν τόσες φάσεις αφενός και αφετέρου να έχουμε μια μέθοδο πιο διαφοροποιημένη Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο γιατί και η Κομισιόν είναι στη διάθεσή μας σήμερα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Φίλιπ Τζεν από την ε, μονάδα ε, το, της, ε, των μηχαν, της μηχανοκίνητης βιομηχανίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, σε ένα σεμινάριο που έλαβε χώρα πριν από λίγο καιρό ε, αναφερθήκαμε ενδελεχώς και ενεκτάσει σε αυτά τα θέματα ε, και νομίζω ότι αντιμετωπίσαμε ακόμα και κάποια ερωτήματα τα οποία είχαν προέλθει από τους βουλευτές Επιτροπής σας εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύουμε ότι πρέπει να επισύρουμε την προσοχή ε, σας ε, στο γεγονός ότι η πρόταση θα πρέπει να δοθεί επίσης και υπό το πρίσμα των τροποποιήσεων που θα λάβουν χώρα και στο τομέα των ελαστικών. Ε, το 12 θα τεθούν σε ισχύ νέες οριακές τιμές όσον αφορά τα ελαστικά και επίσης ε, στην σήμανση θα γίνεται λόγος και στην ενεργειακή απόδοση και στο επίπεδο ε, θορύβου. Βεβαίως δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα ποια θα είναι η επίπτωση στους καταναλωτές, μπορούμε να το φανταστούμε όμως το Νοέμβριο του 2012 ε, θα αρχίσει να εφαρμόζεται το σύστημα της σήμανσης και θα δούμε ε, πώς θα επηρεάσει, ελπίζουμε θετικά βέβαια, τους ε, καταναλωτές και την επιλογή τους. Θα υπάρξει και σήμανση όσον αφορά τον θόρυβο, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι η επίπτωση αυτής της σήμανσης στους καταναλωτές και την επιλογή τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Θόρυβος και μεταφορές. Είναι θέματα που τα συζητήσαμε και με τον Επίτροπο. Ορισμένε φορές ε, πάμε ψάχνοντας για να δούμε τις επιπτώσεις στην υγεία, για παράδειγμα, στο θόρυβο. Στην δική μου πόλη το πρόβλημά μας είναι τα τραμ και τα τρένα. Οπότε έχουμε θόρυβο και από τις ράγες και από το κινητήρα. Το θέμα λοιπόν είναι πώς επηρεάζεται η υγεία από τις πιο διαφορετικές πηγές θορύβων και ποια είναι η κατανομή της επίδρασης αυτής. Α, κάποια ομιλήτρια που δεν είδα η κυρία Μόκενχάιτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε κάτι συγκεκριμένο. Μιλάμε για την χορύπανση που οφείλεται στο χήματα. Όλοι νιώθουμε την ενόχληση από την ηχορύπανση στις πόλεις. Από την άλλη μεριά μιλάμε για τα καινούργια οχήματα. Μήπως θα έπρεπε να μιλήσουμε και για τα μεταχειρισμένα οχήματα. Περί τίνος πρόκειται δηλαδή. Όταν τα οχήματα πολλούνται και αρχίζουν και κυκλοφορούν στην αγορά, έχουν κάποια πιστοποίηση. Όμως, λίγα χρόνια αργότερα, κατά τον τεχνικό έλεγχο διαπιστώνουμε ότι δεν είναι πάντα σίγουρο ότι τα οχήματα αυτά ανταποκρίνονται ε, στα όρια η χορύπανση, γιατί δεν ξέρουμε ποια ακριβώ είναι αυτά τα όρια η χορύπανση που πρέπει να εφαρμόζονται στα μεταχειρισμένα οχήματα. Εφόσον λοιπόν δεν γνωρίζουμε τα δεδομένα της πιστοποίησης, 92 δεσιμπέλη είναι στη Λιθουανία. Αυτόματα φαίνεται πως το επίπεδο της συγχωρήπανσης μπορεί να είναι μεγαλύτερο, ψηλότερο. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ε, ρωτήσω, μήπως θα έπρεπε να προτείνουμε τη δημιουργία μιας κοινή βάσης δεδομένων όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των οχημάτων αυτών για να ξέρουμε ποια είναι τα όρια της συγχωρήπανσης που επιτρέπεται από αυτά. Όσον αφορά τη σήμανση, έθεσα το ερώτημα στον ε, εισηγητή. Αν έχω εγώ ε, έχω την ε, δυνατότητα να με ένα όχημα, δεν θα πρέπει ούτως άλλως να τηρώ τις ε, τιμές που αντιστοιχούν σε αυτόν τον τύπο. Γιατί χρειάζεται πλέον σήμανση. Εν πάση περιπτώσει, να δώσω το λόγο στον κύριο Ούσκι για να μα εξηγήσει, εάν όντω έτσι έχουν τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα την ερώτησή σας για τον τύπο οχημάτων. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι για παράδειγμα ένα μικρό λεωφορείο έχει διαφορετικές προδιαγραφές ε, να τηρήσει από ότι ένα φορτηγό ή ένα αυτοκίνητο σπορ. Η ταξινόμηση της Επιτροπής και η δική μου περιλαμβάνουν αυτές τις διάφορες τιμές. Οι συνάδελφοι έκαναν μερικές ε, ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση Μέρκης. Α, δεν είναι εδώ. Η πρότασή μου είναι να επανέλθουμε σε αρχικές μεθόδους δοκιμών που εφαρμόζονται εδώ και 20 χρόνια. Θα ήταν δύσκολο να εφαρμόσουμε νέες μεθόδους ε, ελέγχου. Οι Γερμανοί είπαν ότι θα μπορούσαμε να δεχθούμε νέες μεθόδους δοκιμών. Για παράδειγμα, να αυξήσουμε την επιτάχυνση από 2 σε 3 μέτρα ανά του τετράγωνο. Είναι σαφές το μήνυμα. Νομίζω ότι αν περιοριστούμε στην αρχική πρόταση θα ήταν πιο θετικό. Όπως είπε και ο Χόλγεν Κράμερ, συμφωνώ 100% με τις εξηγήσει που μας έκαναν οι πράσινοι. Πρέπει να έχουμε πλατιά πρόπτικη. Από ό,τι ξέρω, ο χρόνος έρευνας και ανάπτυξης ενός νέου κινητήρα είναι 8 με 12 χρόνια. Αν είμαστε φιλόδοξοι, πολύ μας αρέσει η λέξη αυτή φιλόδοξη στην Επιτροπή μας, Πρέπει φυσικά να δείξουμε και στην αυτοκινητοβιομηχανία προ τα που πρέπει να πάει. Φυσικά να υπάρξει μελέτη επιπτώσεων μετά την τρίτη φάση, βεβαίω. Τα ηλεκτρικά οχήματα δεν είναι θέμα για την Επιτροπή μας. Πρέπει να συζητήσουμε αν θα πρέπει να αυξήσουμε τεχνητά τον ήχο των ηλεκτρικών οχημάτων για λόγους ασφάλειας. Νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα Weisberger και, και Ίμκο. Περισσότερο αρμοδιότητα δική τους είναι πιστεύω, διότι για την προστασία της δημόσιας υγείας δεν είναι αναγκαίο να αυξήσουμε τεχνητά τον ήχο που παράγουν τα ηλεκτρικά οχήματα. Για την ερώτηση των πρατίνων είναι λιγότερο φιλόδοξη η πρότασή μου. Αλλά κοιτάξτε, άλλοι μου λένε ότι πρέπει να είμαι πιο φιλόδοξος, άλλοι να είμαι πιο ρεαλιστής. Πιστέψτε με συνάδελφοι, Προσπάθησα να σας υποβάλω μια έκθεση που να συνδυάζει τις διάφορες απόψεις. Δεν είμαι σίγουρος ότι κάθε τροπολογία θα έπρεπε να είναι ακριβώς έτσι, ότι αυτή ήταν η βέλτιστη διατύπωση. Αλλά προσπάθησα να συνδυάσω και να λάβω υπόψη τις απόψεις όλων των σκιωδών εισηγητών και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Υπόθηκε για την διαχείριση της κυκλοφορίας των οχημάτων. Ότι αυτό θα αυξήσει τη δυνατότητα χρήσης των αστικών υποδομών. Κοιτάξτε, ένα φορτηγό μπορεί να κάνει το θόρυβο που κάνουν 20 αυτοκίνητα. Άρα Εάν περιορίσουμε την κυκλοφορία στο κέντρο των πόλεων μα, αυτό θα βοηθούσε τη δημόσια υγεία, θα έσωζε σε τελευταία ανάλυση και ζωή. Να καταργήσουμε την πρώτη φάση. Ορισμένοι είπαν το αντίθετο. Πιστεύω ότι μια καλή συμβαστική πρόταση θα ήταν τέσσερι φάσει ε, που να αρχίσουν να εισάγονται ω το πιο σύντομα. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στην περαιτέρω επικοδομητική συνεργασία. Ευχαριστώ, Μύρο Ούτσκι, λέει ο πρόεδρο. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών Ιουνίου 12 το μεσημέρι. Για τι τροπολογίε, θα ψηφίσουμε στι 20-21 Ιουνίου στην Επιτροπή μα, Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στι 10 Ιουλίου και κατά πάσα πιθανότητα στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου 2012 θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια το κείμενο αυτό. Αυτό σημαίνει ότι για δεύτερη ανάγνωση θα είχαμε επαρκή χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Τους ομιλητές. Επόμενο θέμα της μερίσιας διάταξης, μερίσιας διάταξης, το 5, δημόσιες προμήθειες. Η συγκήτρια Όσα Και τη δίνω Κατά προτεραιότητα το λόγο. Η οδηγία αυτή για τις δημόσιες προμήθειες είναι πολύ σημαντική για την Επιτροπή. Όπως ξέρετε, οι δημόσιες προμήθειες είναι 18% του ΑΕΠ, πολλά εκατομμύρια εργάζονται για την ε, ικανοποίηση των ε, δημοσίων προμηθειών. Εάν θέλουμε λοιπόν να εφαρμόσουμε τους στόχους της συνθήκη και του Ευρώπη 2020, οι δημόσιες προμήθειες πρέπει να χρησιμοποιηθούν με έναν τρόπο που να βοηθήσει την αηφόρο ανάπτυξη. Η δική μου αντίληψη είναι ότι η κοινοτική νομοθεσία θα μπορούσε να βελτιωθεί ούτω ώστε να, να καταστεί πιο εύκολο στι δημόσιε αρχέ να αναλαμβάνουν τι ευθύνε του. Πολλοί από του κανόνε θέτουν φραγμού αντί να διευκολύνουν την ε, χορήγηση των ε, δημοσίων ε, συμβάσεων. Ως Επιτροπή Περιβάλλοντος πρέπει να στοχεύσουμε την έκθεσή μας σε αυτά ακριβώς τα ερωτήματα. Προτείνω να επιχειρήσουμε να βελτιώσουμε τη δυνατότητα για να λαμβάνεται υπόψη ο πλήρης κύκλος ζωής μιας υπηρεσίας αγαθού, καθώς και οι κοινωνικές και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις πρέπει οπωσδήποτε η διαδικασία παραγωγής να είναι βιώσιμη και να γίνεται με ίση αμοιβή για ίση εργασία. Οι δημόσιες αρχές που αγοράζουν αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες πρέπει να φροντίζουν να έχουν την καλύτερη τιμή, αλλά να έχουν και την καλύτερη κοινωνική και περιβαλλοντική επίπτωση. Αυτό πρέπει να καθορίζεται εκ των προτέρων για να μην υπάρξει διαφθορά κατά την χορήγηση των συμβολέων. Είναι σημαντική αρχή αυτή της δημοκρατίας Δηλαδή να αποφασίζουμε τοπικά τι προϊόντα θέλετε να αγοράσετε και από πού και υπηρεσίες. Είναι σημαντικό επίσης για την ε, χρηστή διαχείριση των δημοσίων πόρων. Πολλές ε, επικρίσεις έχουν γίνει κατά αυτής της Επιτροπής γιατί περιορίζει διαφόρους ε, τρόπους σήμανσης. Επιχείρησα να επιλύσω το πρόβλημα αυτό μιλώντας περισσότερο για πρότυπα που θα πρέπει να τα ελέγχουν τρίτη Πρέπει να λύσουμε με σωστό τρόπο το πρόβλημα αυτό. Η σήμανση είναι σημαντικό στην αγορά, βοηθάει να προωθήσουμε αϊφόρο παραγωγή και ελπίζω να υποστηριχθεί ευρέως η λύση που επέλεξα. Η αλλαγή στην οδηγία που προτείνει η Επιτροπή επίσης εξετάζει πως μια σειρά δημόσιες αρχές παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες δημόσιες αρχές, για παράδειγμα απόβλητα θα έπρεπε οι δημόσιες αρχές να μπορούν να συνεργάζονται για την ε, κατεργασία αποβλήτων, παροχή ε, ίδρευσης. Όταν πρόκειται για υπεργολαβίες είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχουν συνθήκες στην πολιτική δημοσίων προμηθειών που να περιορίζουν τον αριθμό των υπεργολάβων ούτως ώστε το συμβόλαιο να εκτελείται με τον τρόπο με τον οποίο συμφωνήθηκε και να αυξάνει την ανταγωνιστικότητα. Μια τελευταία τροπολογία λέει ότι η δημόσια αρχή, η αναθέτουσα αρχή όταν αγοράζει μια κοινωνική υπηρεσία μπορεί να, να της αποφέρει και κέρδος. Βέβαια, οποιοδήποτε τέτοιο κέρδος προκύπτει θα έπρεπε να επανεπενδύεται σε δημόσιους στόχους, υγεία, παιδεία κτλ. Ελπίζω λοιπόν τροπολογίες αυτές να εγκριθούν από την Επιτροπή για να επιτύχουμε μια σωστή ευρεία βάση συμβασμού. Ελπίζω οι συνάδελφοι να υποβάλουν τροπολογίες και προσβλέπω στην ε, συνεργασία με τους συναδέλφους και στη λήψη υπόψη των απόψεων άλλων. Ευχαριστώ. Περνάμε στους σκιώδες ηγητές. Πρώτος ο συνάδελφος Μύροσλαπ Μικολάζιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι, ευχαριστώ και την εισηγήτρια Προετοίμασα γραπτά κάποιες απόψεις τις οποίες θα ήθελα να σας κοινοποιήσω και γιατί θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Συμφωνώ απολύτως με την εισηγήτρια ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και για την Επιτροπή μας και για άλλες επιτροπές. Είναι πολύ ελκυστικό, είναι πολύ σεξι λέει ο αυτό το θέμα αυτό. Ε, να μοιραστώ λοιπόν κάποιες σκέψεις ε, μαζί σας. Η σύλληψη δημόσιων συμβάσεων είναι πολύ σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης και βοηθάει στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς μπορεί να καλύψει ανάγκες σε υπηρεσίες, αγαθά ε, και υποδομές, ε, έτσι ώστε να ε, είναι οι δημόσιες συμβάσεις όσο γίνεται πιο αποτελεσματικές και να καταλήξουν σε βιώσιμη και διαρκή ανάπτυξη, οπωσδήποτε θα πρέπει να τεθούν κάποιες προϋποθέσεις. Η συγγήτρια Άσα Βέστλουντ ορθώς αναφέρει ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις και, και τα οποία αφορούν την οικονομία και το περιβάλλον. Αυτά τα στοιχεία ορθώς αναφέρονται στο προσχέδιο της έκθεσης πιστεύω ότι θα πρέπει να απλουστευθούν τα πράγματα, ε, αλλά ταυτόχρονος θα πρέπει να αναπτυχθούν, να αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό των δημοσίων συμβάσεων μέσω τροποποίηση των κανόνων. Σε συνεργασία με καινοτόμα και βιώσιμα κριτήρια, τα οποία θα είναι ταυτόσιμα με αυτά της στρατηγικής 2020, θα πρέπει να καλύψουμε ε, φιλόδοξους στόχους ε, για την κοινωνική η συνοχή, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή, την εκπαίδευση, έτσι όπως αυτοί οι στόχοι αναφέρονται ε, στο, 20, στο πρόγραμμα 2020. Ε, Επίσης θα πρέπει να ληφθούν αυτές συγκεκριμένες δράσεις σε εθνικό αλλά και ενωσιακό επίπεδο έτσι ώστε να στηριχτεί η στρατηγική αυτή. Πιστεύω ότι και η καινοτομία και ο ανταγωνισμός θα πρέπει ε, να έχουν έναν νέο προϋπολογισμό. Ε, ελαφρότερο ε, διοικητικό άχθος επίσης ε, όσον αφορά τις αρχές των δημοσίων συμβάσεων. Ε, είναι γεγονός ότι οι τοπικές αρχές, ε, είτε είναι δήμοι, κοινότητες, περιφέρειες, θα πρέπει να προχωρούν στις δημόσιες συμβάσεις έχοντας και την απαραίτητη πολιτική προστασίας πιστεύω ότι θα πρέπει το κριτήριο της ελάχιστης ε, τιμής, ε, της μικρότερης τιμής ε, να καταργηθεί έτσι ώστε οι τοπικές αρχές να είναι αυτές οι οποίες να μπορούν να αξιολογήσουν μια πρόταση και μια προσφορά σύμφωνα και με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, κοινωνικό αντίκτυπο κλπ. Ε, στον τομέα της ε, ασφάλειας, της υγείας ε, και των τροφίμων θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί πρόκειται για συμβάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για τους τελικούς αποδέκτες λαμβάνοντας υπόψη ε, τον, ε, τον, ε, το, τον λαμβάνουμε υπόψη τον κύκλο ζωής των αγαθών μπορεί να μας βοηθήσει και βεβαίως πάντα λαμβάνοντας υπόψη και την καινοτομία. Τέλος να πω ότι στηρίζω τη θέση της εισηγητρίας ότι η νέα οδηγία δεν θα πρέπει να δυναμητίζει την δυνατότητα των τοπικών αρχών να ε, κάνουν δημόσιες συμβάσεις για κοινά αγαθά όπως είναι το νερό ας πούμε. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ανώνη εξ ονόματος ε, της Άλντε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Διαβάζω την ανάλυση του συναδέλφου Μάντες ε, που είναι σκιώδης και δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ. Ε, ευχαριστώ την εισηγήτρια για την σκληρή και δύσκολη ε, εργασία της. Ε, η ομάδα ALDE δέχεται θετικά την πρόταση της Επιτροπής για μια νέα οδηγία για τη σύνοψη δημοσίων συμβάσεων. Η βελτίωση της εσωτερικής αγοράς και της αποτελεσματικότητας των δημοσίων συμβάσεων αποτελεί, αποτελούν μάλλον συγκεκριμένες προτεραιότητες για μας. Θα πρέπει δε να παίξουν σημαντικό ρόλο στρατηγική στρατηγική 20, Ευρώπη 2020 σαν ένα από τα κυριότερα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην αγορά έτσι ώστε να υπάρξει ευφυής και ολοκληρωμένη ανάπτυξη με σωστή χρήση των δημοσίων πόρων. Κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά το προσχέδιο της έκθεσης. Ε, οι αρχές ε, οι οποίες ε, δίνουν την τελική άδεια για τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Κριτήριο, ε, ε, κριτήρια χωρίς αυτό όμως να είναι ε, πάντοτε απαραίτητο. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα πρέπει να έχουν και αυτές την ευκαιρία να συμμετέχουν στις δημόσιες συμβάσεις. Επίσης οι εταιρείε αυτές θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα διεύρυνσης των δραστηριοτήτων τους και όχι περιορισμού η συγκήτρια μέσω τροπολογιών της ε, προτείνει κάποιες τροποποιήσεις όσον αφορά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Αυτές οι τροπολογίες ε, βρίσκουν σύμφωνη την ε, ομάδα των φιλελευθέρων. Επίσης, ε, η χρήση των ε, ε, αρχών μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη ταυτοποίηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων που θα πρέπει να έχουν κατά νου και να εφαρμόζουν αυτοί οι οποίοι τελικά συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις. Ευχαριστούμε πολύ για την εισηγήτρια για την εργασία της. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλα είναι θετικά εδώ. Οι βασικές ιδέες από πλευρά της Επιτροπής Περιβάλλοντος πρέπει να ακουστούν. Επέκταση του ορισμού των πιο εποφελών διαδικασιών που περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές είναι μια πολύ θετική προσθήκη. Βέβαια δεν είναι όλα στο χέρι μας. Ένα από το βασικό πρόβλημα των δημόσιων συμβάσεων είναι ότι είναι πολύ περίπλοκες για τις περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεν εκμεταλλεύονται πάντα τις δυνατότητες που έχουν στη διάθεσή τους, ώστε όντω να συμπεριλάβουν τέτοιες περιβαλλοντικές η κοινωνικές προδιαγραφές. Άρα το βασικό είναι απλοποίηση. Αυτά που προτείνει η είναι θετικά. Ένα ορισμός που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ είναι αυτό στον οποίο έχουν καταλήξει και οι Ηνωμένε Πολιτείε που λένε ότι δεν θα πρέπει να είναι κάτι δογματικό, μια δογματική βεβαρημένη ιδεολογικά αγορά, αλλά θα πρέπει να είναι κάτι ανοιχτό σε όλου. Όταν έχουμε να κάνουμε με την αγορά τροφίμων. Ας δούμε τι έχει γίνει στι Ηνωμένε Πολιτείε. Πολλέ πολιτείες, στι Ηνωμένε Πολιτείες, έχουν τέτοιες ε, ζητάνε δημόσιε προσφέρε και πρέπει να δούνε ποιο ε, υπακούει στα κριτήρια και κοιτάνε αν υπάρχει διαφορά πάνω από 5% μεταξύ δύο προσφερόντων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ε, το κοιτάξουν αλλιώς, αλλά αν διαφορά είναι κάτω από 5% τότε δίνουν την προσφορά στον πιο κοντά στην ε, πολιτεία ε, προσφέροντα. Ας δούμε λοιπόν και εμείς αυτή τη δυνατότητα. Όπως προτείνει και η συγγήτρια, προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε και στοιχεία όπως είναι η προστασία των ζώων και άλλες προδιαγραφές. Όταν έχουμε να κάνουμε με δημόσιες συμβάσεις για την αγορά κρέατος, τότε Βέβαια, το θέμα αυτό έχει μεγάλη σημασία το να το βάλουμε, όμως εδώ δεν ξέρω, σε αυτήν την γνωμοδότηση δηλαδή δεν ξέρω. Κάτι άλλο είναι νέες δυνατότητες για τις δημόσιες αρχές προκειμένου να αγοράζουν υπηρεσίες. Δεν είναι μια συνήθις διαδικασία, γιατί κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για μια σύμβαση Υπάρχει βέβαια ανταγωνισμός. Αυτό που είναι σημαντικό είναι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές να έχουν τη δυνατότητα να έχουν ευκαιρίες προκειμένου να συμπεριλάβουν και ελάχιστες απαιτήσει περιβαλλοντικές και κοινωνικές που να τις λαμβάνουν υπόψη τους όλοι όσοι υποβάλλουν τις προσφορές τους. Φυσικά δεν μπορείς να προκαταλάβεις ε, τα πράγματα γιατί δεν ξέρεις ποιος πελάτης θέλει τι. Αλλά νομίζω ότι γενικά είναι πολύ καλή πρόταση που έχουμε και θα καταλήξουμε σε μια καλή ε, πρόταση τελικά. Γιατί αυτό που θέλουμε είναι η φόρα ανάπτυξη για όλους. Όταν όμως πέει κανεί να αγοράσει, δεν έχει αυτό στο μυαλό του. Έχει στο μυαλό του να αγοράσει το καλύτερο δυνατό προϊόν στην καλύτερη δυνατόν τιμή. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι να συμπεριληφθούν και περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια σε αυτές τις αγορές. Για να αξίζουν τον κόπο τα λεφτά που δίνουμε. Ευχαριστώ. Julie Βεβαίω ε, συμφωνώ με όλοι ότι πρέπει οι εταιρείε μας να έχουν ε, πολύ περισσότερες ευκαιρίες για να βελτιώσουν ε, την ανταγωνιστικότητά τους αλλά και την συμμόρφωση με τις διάφορες απαιτήσει. 20% του ΑΕΠ ε, είναι σημαντικό ποσοστό, πολύ σημαντικό για όλους. Στην πρόταση της Επιτροπή αναγνωρίζει τις ανησυχίες αυτές και η πρότασή της είναι ιδιαίτερα ευραίος φάσματος, ε, ριζικές αλλαγές, το καλωσορίζω και ισχυρή ε, κίνηση προς περισσότερη ευελιξία και αυτό το καλωσορίζω. Και βεβαίω. ε, μου αρέσει πάρα πολύ το τμήμα της έκθεσης της Κομισιόν που μιλάει για εταιρικέ σχέσεις για την καινοτομία. Συνεργασία για την καινοτομία. Καλό επίση αυτό που λέει πως δεν είναι μόνο ο δεν θα πρέπει υποχρεωτικά ομοιοδότης που θα πρέπει να παίρνει κάθε δημόσια προμήθεια. Πρέπει να καθορίζεται βέβαια σαφώς τα άλλα κριτήρια. Βεβαίω, θα έπρεπε να υποστηριχθεί ιδιαίτερα αυτή η συνεργασία για την καινοτομία. Από περιβαλλοντική άποψη αυτό δεν αναφέρεται παρκώς στη γνωμοδότηση. Νομίζω ότι η γνωμοδότηση επίσης ε, μπαίνει σε χωράφια που δεν είναι δικά της. Ιδιαίτερα αυτό το θέμα για την εργασία και η αναφορά στην Σύμβαση 94 του Παγκοσμίου Γραφείου Οργασίας. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει αλλού αν ε, είναι σχετική με τις δημόσιες προμήθειες. Δεν νομίζω όμως ότι είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Είναι κάτι που θα έπρεπε να το εξετάσει η Επιτροπή Απασχόλησης. Και ως μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης είναι ότι εάν επιχειρήσουν σε οτιδήποτε περιβαλλοντικό θα τους ε, κατακεραυνώναμε. Νομίζω ότι και εμείς πρέπει να το κάνουμε λοιπόν. Να μην μπαίνουμε στα χωράφια τους. Επίσης ο ορισμός οι παραγωγικές διαδικασίες, οι κοινωνικά βιώσιμες παραγωγικές διαδικασίες. Δεν είναι και τόσο σαφές βεβαίως. Πολλές από τις τροπολογίες είναι ταυτόσιμες με αυτές που υπήρξαν στην ΙΜΚΟ. Αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει αυτή η έννοια. Αν δούμε την τροπολογία 11 που προσπαθεί να ορίσει αυτό το θέμα με βάση κριτήρια κύκλου ζωής. Είναι όσο σαφής είναι και η λάσπη. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να εισαγάγουμε ασαφής. Ναι, μεν η πρόθεση είναι αξιέπαινη, δεν την επικρίνω, αλλά στόχος μας πρέπει να είναι όλοι στην διαδικασία του κύκλου παραγωγής πληρούν αυτά τα οποία θα αποφασίσουμε. Δεν είναι εύκολο να το ορίσουμε. Εάν δεν υπάρχει σχέση με το θέμα του ε, συμβολέου, θα μπορούσαμε να έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Θα μπορούσε να σταματήσει η όλη διαδικασία δημοσίων προμηθειών γιατί θα μπορούσε να αμφισβητηθεί οποιοδήποτε συμβόλαιο. Από πού προέρχεται αυτή η έννοια και ποια είναι η νομική της βάση. Οπότε, οπότε πρόθεση βεβαίως κάθε κειμένου είναι να μειωθεί η υπερητή γραφειοκρατία αλλά τελικά όλες οι προτάσεις που γίνονται πιστεύω πως πηγαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο στην Επιτροπή την ευκαιρία να πάρει το λόγο. Θέλει κανείς από την Επιτροπή το λόγο. Παρακαλώ. Διάνο από την Γενική Διεύθυνση Αγοράς. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και, για... και ευχαριστώ και όλους για τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε. Έχω ένα μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απομακρυνθείτε λίγο, λέει ο Πρόεδρος, από το μικρόφωνο, γιατί γίνεται μικροφωνισμός, δεν ακούγεστε καλά. Ένα γενικό μήνυμα θέλω να σας μεταφέρω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι ότι οποιαδήποτε παρατέρω πρόταση ή οτιδήποτε άλλο έχετε να προτείνετε πρέπει να βασίζεται στις συνθήκες. Ιδιαίτερα το θέμα αυτό της μη διάκρισης, οποιαδήποτε τροπολογία δηλαδή, δεν θα πρέπει να οδηγεί σε διακρίσεις. Επίσης θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι δεν πρέπει να προσθέσουμε διοικητικό άχθος. Ακούσαμε πολλά για ε, τη, τους ανάδοχους, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ο φόρτος εργασίας. Η συγγήτρια τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. πίστευα και εγώ ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για να καταλήξουμε σε ικανοποιητικέ λύσεις. Αυτό το οποίο επανέρχεται συνέχεια είναι το πώς εκείνοι οι οποίοι αποφασίζουν θα μπορέσουν να δουν και την καλύτερο και το εκλογικό του σώμα και να έχουν την αίσθηση ότι αυτό ακριβώς αποφασίζουν και όχι ότι έρχεται κάποιος από πάνω και τους επιβάλλει τις αποφάσεις τους. Το πιο σημαντικό όταν έχουμε διάφορους που υποβάλλουν προσφορές από ολόκληρη την Ευρώπη, το πιο σημαντικό είναι να καταφέρεις να βρεις το δρόμο σου και να επιλέξεις τελικά αυτό που πραγματικά θέλεις. Αυτό το οποίο αγοράζετε τοπικά λοιπόν πρέπει να αποφασίζετε και τοπικά. Αυτό είναι το κύριο κριτήριο. Και πιστεύω ότι υπάρχει εδώ μεγάλος βαθμός συνένεσης. Αν ρωτήσετε τους ανθρώπους στην Ευρώπη και τους πολιτικούς, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει συνένεση. Τώρα για τα διάφορα επιμέρους θέματα. Εγώ προσπάθησα να περιοριστώ εκεί που εμείς έχουμε κάποια αρμοδιότητα. Δημόσια υγεία σε ένα βαθμό, Όντω είναι ένα θέμα που πρέπει να αναφέρεται στην ε, έκθεσή μας, ε, όπω η αγορά εργασίας. Βέβαια, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να έχει μια διαφορετική άποψη. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση αυτή, γιατί υπάρχουν χιλιάδες ε, δήμαρχοι, για παράδειγμα, και δημοτικοί σύμβουλοι που τους αφορά, και πρέπει λοιπόν να είμαστε ευέλικτοι όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες τους διαγωνισμούς, αλλά μας ενδιαφέρει βεβαίως να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και τα περιβαλλοντικά κριτήρια. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προπαρασκευάσουμε την οδό και για να το κάνουμε αυτό προθεσμία υποβολή τροπολογιών 7 Ιουνίου 12 η ώρα το μεσημέρι παρακαλώ. Η τροπολογία θα γίνει πριν, η ψηφοφορία συγγνώμη, θα γίνει 10 Ιουλίου την ΙΜΚΟ που είναι επί του αρμόδια. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου και κατά πάσα πιθανότητα το Δεκέμβριο θα περάσει σε πρώτη ανάγνωση στην Ολομέλεια. Όπου και θα ψηφιστεί. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ε, παρευρισκόμενους. Τα άλλα δύο σημεία της ημερής διάταξης είχα ανακοινώσει στην αρχή τα 6 και 7 ότι αναβάλλονται για την επόμενη συνεδρίασή μας. Οι συντονιστέ, παρακαλώ να είναι εδώ αύριο στι 9 για συνεδρίαση των συντονιστών. Όλοι οι άλλοι παρακαλώ ε, να είναι 10 ακριβώς εδώ γιατί θα αρχίσει η ψηφοφορία. Παρακαλώ να φέρετε τις κάρτες ψηφοφορία για να μπορέσουμε να κάνουμε τι ψηφοφορίε απρόσκοπτα. Καλό βράδυ.